Can I bring the meeting to... Παρακαλώ να αρχίσουμε. Καταρχήν να σας πληροφορήσω τι συζήτησαν οι συντονιστές. Οι συντονιστές αποφάσισαν να μην κάνουν τίποτε για τον ορισμό εισηγητών για ορισμένες τροποποιήσεις συμβάσεων αλλά να γράψουν, γραφτούν τρεις γνωμοδοτήσεις. Πρώτον, η τροποποιημένη πρόταση κάνουν για κανονισμό για κοινέ ρήτρε, για το Περιφερειακό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής και άλλα όπως την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αλία. Οι πράσινοι το αναλαμβάνουν. Δεύτερη, πρόταση κανονισμού για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων η φιλελεύθερη και τρίτη γνωμοδότηση για την αναγνώριση των βελτίστων πρακτικών στην ανάπτυξη της υπαίθρου είναι αρμόδια η Επιτροπή Γεωργίας, έχει και ένα στοιχείο τουρισμού και η Γκούε θα το αναλάβει αυτό. Η ακρόαση στις 29 Μαΐου για τα δικαιώματα των επιβατών θα αναβληθεί για το Σεπτέμβριο για το κόστος της μη Ευρώπης στις μεταφορές αποφασίσανε να γίνει έκθεση για τη συμβολή της ΜΕΤΑΦ στις στρατηγικές πρωτοβουλίες κατόπιν επιστολής του Προέδρου της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά να γραφτεί επιστολή μέχρι τις 15 Μαΐου το Γενικό Γραμματέα για την εσωτερική αγορά, άλλη επιστολή του κ. Χάρμπορ για ψήφισμα για την κυβερνοασφάλεια στην Ένωση. Θα γράψω επιστολή στον πρόεδρο της ΙΜΚΟ για αυτό το θέμα και ό,τι σχετίζεται με τις μεταφορές. Προφορική ερώτηση για την οδική ασφάλεια αποφασίσαμε να ζητήσουμε να συμπεριληφθεί στην Ολομέλεια του Ιουνίου και αν έχουν οι ομάδες σχόλια να τις υποβάλουν στη γραμματεία μέχρι τις 17 Μαΐου. The decision was to invite the Commission to a future committee meeting. Αποφασίσαμε για την ευθυγράμμιση να ακούσουμε και περαιτέρω προτάσεις για την επιτροπολογία σημειώσαμε την επιστολή παριθμών 9 αυτά είπαν οι συντονιστές σας κατευχαριστώ είναι όλοι ικανοποιημένοι ο κύριος Μπράντπορν ευχαριστώ πρόεδρε Μιλήσατε για την ακρόαση για τα δικαιώματα των επιβατών που το συζήτησαν οι συντονιστές. Από ό,τι κατάλαβα, η, τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές είχαμε πει ότι θα συνόδευαν το γενικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των επιβατών γενικώ, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα καινούριο μάθατε μήπως ή κανείς άλλος έμαθε αν θα υπάρξει αυτή η προσθήκη. Δεν ξέρω τίποτα σχετικά. Η ακρόαση αυτή αφορά συγκεκριμένα την τροποποίηση στον κανονισμό 261. Μπορώ να ρωτήσω την Κομισιόν ή μπορεί και να μας το πουν γραπτός αν προβλέπετε τίποτα συγκεκριμένο για τις αερομεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών. Μάλιστα. Λοιπόν, ψηφοφορίες. Πρώτον δοκιμή, ηλεκτρονική δοκιμή παρακαλώ, άρχεται η εικονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε. Ένας παραπάνω του ΕΛΚ. κύριε Γκρός. Για διαλέξτε κάποιον από τους δικούς σας που να μην ψηφίσει. Μάλιστα. Ο Μαρινέσκου είναι εδώ, ναι. Για να αρχίσει την έκθεσή του βέβαια γιατί ξέρω ότι υπήρξαν ορισμένα προβλήματα στις συγκοινωνίες. Μου είχαν πει ότι θα μπορεί να αργούσατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας πληροφορήσατε εν καιρός, αν και ήρθατε. Λοιπόν, είναι έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ, αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Ε, εισηγητής, όπως σας είπα, είναι ο κύριος Μαρινέσκου. Έτοιμοι, φύγαμε. Μετά την παράγραφο 1, ίντα 1, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ίντα 2, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 9. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 5 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 της επιτροπή Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 της ίδιας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 13 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται άρα η 12 καταπίπτει 4 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 επιτροπής απασχόληση υπέρ α όχι έχει καταπέσει έχει καταπέσει 18 τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα του 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε πέρας εγκρίνεται 24 υπέρ κατά για την 24 έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσετε πέρας τη ψηφοφορίας απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 κατά τμήματα πρώτο τμήμα μέχρι όλο το κείμενο με την εξαίρεση το κόστος των εκπομπών ε, άνθρακα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το δεύτερο τμήμα με τις λέξεις αυτές υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 επιτροπή απασχόληση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 της ίδιας επιτροπής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 της επιτροπής απασχόληση, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 5 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την τα 5 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίσετε πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 απασχόληση υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 23 της Επιτροπής Απασχόλησης άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζεται Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. Είναι τα τρία υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 14 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 17 της ίδιας Επιτροπής υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο. Ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 17 της Επιτροπής Απασχόλησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζετε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 18 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 της ίδιας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε έλεγχο για τη 41 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 22 προς 20 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τοπολογία 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 52 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίντα 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 μπένιον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές έλεγχος νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία Α ψηφίσατε όλοι πέρασε τι ψηφοφορίε. πέρασε εγκρίνεται 23 προς 21 καλά κάνουμε και τσεκάρουμε τροπολογία 1 φώστερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά, αποχές, έλεγχος, αν και νομίζω ότι απορρίφθηκε. Για την τροπολογία 2, Λίχτεμπεργκερ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3, Φώστερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και β της Επιτροπής Απασχόλησης, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Ψηφίζουμε μάλλον ηλεκτρονικά. Ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κανείς καμία αρνητική ψήφο, ψήφος. Τρεις ε, αποχές. Ευχαριστήρια κύριε Μαρινέσκου. Προχωρούμε. Σχέδιο σύστασης για την πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη τη συμφωνία για ορισμένε διαστάσει ε, των υπερπαρχή περιοριζών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη κυβέρνηση τη Δημοκρατική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Σρι Λάγκα. Μία ψηφοφορία με τον κύριο Σαρβανό. Ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 43 υπέρ, καμιά ψήφος κατά, ούτε αποχή, δεκτό. Προχωρούμε. Τροποποίηση του κανονισμού είναι ε, του Συμβουλίου για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορισμένης κατηγορίας οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων και του κανονισμού για τις δημόσιες συμβάσεις. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, κάποιες μέσω του εισηγητή. Η τρία είναι ίδια όπως η δέκα. Μαζί μπορούμε να τις ψηφίσουμε αν θέλετε. Ωραία. πρέπει να πάμε στην αιτιολογική σκέψη 11 χωριστά, γιατί μια καταπίπτει. Άρθρο 1, 3 ε, και 10 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Προχωρούμε στην αιτιολογική σκέψη 11, τροπολογία 2 του συγητή, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Αυτό σημαίνει ότι 7 καταπίπτει. Τώρα, η τροπολογία 9 στην ιδιολογική σκέψη 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Και για πρώτη φορά στην πολιτική μου σταδιοδρομία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πέρασα ε, έκθεση με ε, ψηφοφορία ομόφωνη. 44 υπέρ, χωρίς κατά, χωρίς αποχές. Μου πέρασε, χρειάστηκαν 25 χρόνια, αλλά το κατάφερα. Ωραία. Τώρα περιμένουμε να πάει η ώρα 10 για να αρχίσει η ακρόαση. Επειδή είσαστε τόσο καλοί, ταχύτατοι, θα σας δώσω μισή ώρα διάλειμμα μέχρι τις 10. Συνάδελφοι, ελάτε λίγο πριν από τις 10 για να αρχίσουμε στην ώρα μας και να εκμεταλλευτούμε το χρόνο 100%. Ευχαριστώ.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 Ladies and gentlemen, can I ask you... Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Everybody's down there. Yeah. Okay. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω γιατί έγινε συσκότηση από τώρα. Συνεχίζουμε όμως. Θα ήθελα να αρχίσω αυτή την πρώτη συνεδρία του δημόσια ακρόαση για την τέταρτη δέσμη μέτρων για το σιδηρόδρομο. Σήμερα το πρωί θα εξετάσουμε το άνοιγμα των αγορών, των εθνικών αγορών για τους επιβάτες και για μια καλύτερη διακυβέρνηση για τους σιδηροδρόμους μέχρι τις 12.30. Ελπίζω να προλάβουμε να πάρουμε τις ερωτήσεις μέχρι τις 11.30. Το απόγευμα θα εξετάσουμε τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια και τις αρμοδιότητες του ΕΟΣ, του Εθνικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι διότι καταφέραμε να έχουμε 16, 13, 13, συγγνώμη, 13 ομιλητές για την ακρόαση αυτή μέσα στην ημέρα, πρωί και απόγευμα. Είχα πάνω από 30 αιτήματα από, διάφορες οργαν... από διάφορους οργανισμούς που ήθελαν να συμμετέχουν και να μας μιλήσουν σε αυτή την ακρόαση. Δυστυχώς όμως δεν μπορούσαμε να ε, προσφέρουμε το λόγο σε 30 ομιλητές, ακόμα και με την καλύτερη θέληση. Ζητώ συγγνώμη αν δεν σας συμπεριέλαβα, δεν είναι προσωπικό θέμα αυτό. Έπρεπε όμως να μπορέσουμε να έχουμε ένα μέγεθος διαχειρίσιμο. Ένα πρόβλημα ήταν ότι οι περισσότεροι ήθελαν να μιλήσουν στο πρώτο μέρος της ακρόασης και όχι στη δέσμη μέτρων συνολικά. Αν πιστεύει κάποιος ότι ε, παραγωνίστηκε ο οργανισμός του. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Άλλωστε γνωρίζετε ότι μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τα μέλη, οι περισσότεροι το έχετε κάνει, για να δώσετε τις λεπτομέρειες των απόψεών σας. Αυτή η δέσμη μέτρων είναι πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, σίγουρα εδώ για το Κοινοβούλιο, αλλά και για άλλα κοινοβούλια λόγω της απογοήτευσης ε, που υπήρχε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα και την έλλειψη εσωτερικής αγοράς και ε, πρόβλημα στο άνοιγμα του τομέα των σιδηροδρόμων και της αγοράς τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να μπούμε σε αυτή τη διαφοροποίηση διάκριση εθνικού ευρωπαϊκού, θα ήθελα να πω ότι εμείς εδώ βέβαια υιοθετούμε μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση των σιδηροδρόμων και όχι εθνική. Ένα από τα προβλήματα του παρελθόντος ήταν οι εθνικιστικές απόψεις που επικρατούσαν των πανευρωπαϊκών ή της πανευρωπαϊκής άποψης. Ο πρώτος ομιλητής μας Α, να πω στους ομιλητές ότι θα τηρηθεί αυστηρά το δεκάλεπτο. Θα είμαι αμήλικτος, όπως θα είμαι και με τα μέλη του Κοινοβουλίου αργότερα. Αλλά για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα μην υπερβείτε το δεκάλεπτο. Ε, είχαμε πρόσφατα ακροάσεις όπου οι ομιλητές ε, ξεπερνούσαν το χρονικό περιθώριο και υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, έκκληση. Τηρήστε το δεκάλεπτο. Ο πρώτος μας ομιλητής θα μας μιλήσει για την προοπτική του ε, νέου εισερχόμενου. Είναι διευθύνων Σύμβουλος της Westbahn της Αυστρίας. Δέκα λεπτά, κύριε Φόρστερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας μιλήσω για τη Westbahn, θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες και μετά θα σας μιλήσω για την πορεία της επιχείρησης. Κάποια στοιχεία για την εταιρεία μας την Westbahn. Εμείς ε, έχουμε ε, διαδρομή Βιέννης, Λίντς, Ζάλσμπουργκ, Φραϊλάσινγκ και κάθε ώρα σχεδόν έχουμε εξυπηρέτηση. Είναι 3,16 εκατομμύρια τα ε, σιδηροδρομικά χιλιόμετρα τώρα που προσφέρονται. Είναι υψηλής ποιότητας το σέρβις ε, σε τιμή πάρα πολύ εξυπηρετική, καλή. Έχουμε τέσσερα μπιστρό, δωρεάν Wi-Fi και Και προσπαθήσαμε με την προσφορά μας να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες. Ένα έτος έχουν τα εισιτήρια ε, ισχύ, μπορούν να αλλάξουν όποτε θέλετε, επιστρέφονται αν είναι η κανονική η τιμή και όταν υπάρχει καθυστέρηση, σπάνια πρέπει να πω, τότε ε, υπάρχει ε, μια επιστροφή μείον 25-50% ε, για καθυστερήσεις και χωρίς να κάνει τίποτα αυτομάτως δίνεται ένα κουπόνι. Ποιες είναι οι προσδοκίες που είχαμε πριν μπούμε στην αγορά. Ήταν απλές. Για τους επενδυτές θέλαμε δίκαιες και ισότιμες ευκαιρίες για απόδοση των επενδύσεων ε, θεμητό ανταγωνισμό, δίκαιο ανταγωνισμό από όλες τις πλευρές και συνθήκες χωρίς διακρίσεις. Και δεν θα σας δείξω μόνο την προοπτική του νεοεισερχόμενου στην αγορά, αλλά θα κάνω μια σύντομη περίληψη αυτών που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι θα σας δείξω το φάσμα της απελευθέρωσης με πολύ σαφή τρόπο χωρίς προβλήματα, απλά, γρήγορα πήραμε το πιστοποιητικό ασφαλείας, την άδεια κυκλοφορίας και η έγκριση των οχημάτων που έγινε κυρίως στην Ελβετία γιατί αγοράσαμε ε, ελβετικά, ελβετικούς σειρμούς, ε, ε, δεν είχαν κανένα πρόβλημα, η αποδοχή ήταν συνολική στην Αυστρία Τώρα δεν έχουμε έγκριση για τη Γερμανία. Υπάρχουν εκεί κάποια προβλήματα με την αυτόματη ε, αποδοχή. Τα πρώτα προβλήματα προέκυψαν με τις πρώτες γραμμές και το ε, πρόγραμμα ε, που είχαμε, γιατί εμείς είχαμε πάρα πολύ σαφή σχεδιασμό στην Αυστρία και τα παραδώσαμε στην αρμόδια αρχή και πήραμε το ε, πρώτο μας το ε, πρόγραμμα ε, χρόνος ταξιδίου 2, και 45, 2 ώρες και 45 λεπτά για τη Βιέννη Ζάλσμπουργκ. Ε, μετά ακολουθήθηκε ε, διαδικασία ρυθμιστικού φορέα για την ε, Επιτροπή Ελέγχου Ασφαλείας που κατέληξε στο τρίωρο για το χρόνο ταξιδίου. Εν τω μεταξύ βελτιώθηκε κατά πολύ η κατάσταση, δεν είχαμε δυσκολίες με το δεύτερο πρόγραμμα και με το τρίτο πρόγραμμα για το 2014 ε, δεν υπήρξαν παρεκκλήσεις, αλλά προσθέτω ότι Παντού στον ανταγωνισμό υπάρχει το πρόβλημα ότι ε, πολλές φορές ε, δεν ε, τηρείται απόλυτα το χρονοδιάγραμμα και με βάση το ωριαίο πρόγραμμα θα πρέπει η σειρμή να είναι τέσσερις μέσα στην ώρα κάθε 20 λεπτά και πολλές φορές δημιουργούνται κάποιες συμφορήσεις εκεί. Βασικά όμως δεν υπήρχαν προβλήματα και αν δούμε το ανταγωνιστικό περιβάλλον συνολικότερα, θα πρέπει να πούμε σαφεώς ότι ο ανταγωνισμός διέπεται από το εξής χαρακτηριστικό. Στην Αυστρία απέχουμε πολύ από τον ανταγωνισμό μέσω διαγωνισμών. Το 2010, βάσει νόμου, δόθη η δυνατότητα απευθείας αναθέσεων για ε, υπηρεσίες άνω των 100.000 ευρώ και αυτό εφαρμόστηκε με το σύστημα άμεσ, απευθείας αναθέσεων αναδρομικά από τον Απρίλιο του 2010 από τους Αυστριακούς σιδηροδρόμους. Ε, συνολικά ε, καλύφθηκε μια απόσταση 71 εκατομμυρίων σιδηροδρομικών χιλιόμετρων, που είναι περίπου το 80% ε, των υπηρεσιών που καλύπτουν οι Αυστριακοί σιδηρόδρομοι. Ε, η Βέστμπαν όμω ε, έκανε προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και η απόφαση θα ληφθεί περίπου σε δύο χρόνια. Ε, τώρα υπάρχουν νέες απευθείας αναθέσεις, δηλαδή δεν υπάρχει ε, διαγωνισμός. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε πολύ, ε, λίγο πριν μπούμε στην αγορά, ε, ήταν το εξής στο εθνικό δίκτυο από τους αυστριακούς σιδηροδρόμους ε, έγινε μια προσφορά από 9 ευρώ και μια άλλη στο τομέα του promotion και από το 2005 μέχρι το 2009 ε, υπήρχαν αυξήσεις ε, γύρω στο 3,5% κάθε χρόνο. Από το 2009 μέχρι το 2013 12 λέει εδώ, 13 λέω εγώ. Ε, υπήρξε μία φορά μια αύξηση ε, στα μέσα του 2012. Αν το υπολογίσουμε με βάση την τετραετία, έχουμε πολύ χαμηλότερη μέση αύξηση. Και ε, μετά κάναμε την προσφυγή. βέβαια ένα πράγμα που μας απασχολεί πολύ είναι η υποδομή ε, και η χρέωση για αυτήν. Το 2012 ήταν 4%, περίπου 10%, τώρα 14%, του χρόνου 14%, φέτος 9,8% είναι η ετήσια αύξηση του κόστους υποδομής. Αυτό έχει μεγάλη επίδραση όπως καταλαβαίνετε ε, διότι η υποδομή της Westman επεκτείνεται και είναι ε, περίπου 13 και όχι 10 εκατομμύρια το κόστος αυτό σημαίνει ότι έχουμε απόκληση και πρόσθετη χρέωση ε, αν ληφθεί άλλη απόφαση από εκείνη που έλαβε ο ρυθμιστικός φορέας, που το ελπίζω, τότε θα λυθεί και το πρόβλημα αυτό. Επίσης, πέρα από τη δική μας κουλτούρα προσφοράς, ε, υπάρχει και μία συμφωνία ε, με τους ε, αυστριακούς σιδηροδρόμους που, κάνει την, που έχει μια κάλυψη 80% στο εθνικό δίκτυο. Και για να μην υπερβώ το χρόνο, θα επιταχύνω λίγο. Τώρα, σε λειτουργικό επίπεδο δεν έχουμε προβλήματα. Ε, αντιμετωπίζουμε τα θέματα ε, διακρίσεων. Στο παρελθόν όμως αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα ε, για να ανταποκριθούμε στα... στις προδιαγραφές του ρυθμιστικού φορέα. Ε, τώρα έχουμε... Στην ε, μας είχαν ε, αρνηθεί την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Τώρα ε, έχουμε ε, ε, παλιά ε, είχαμε, μας είχαν δώσει ένα πολύ μικρό χώρο για την Westband, δηλαδή στο, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς που δυσκόλευε ακόμα και τις κινήσεις μας εκεί. Τώρα λύθηκε το θέμα αυτό. Επίσης μπορούμε τις πληροφορίες μας τώρα να τις δίνουμε απρόσκοπτα. Ε, θέλουμε επίσης να έχουμε ενημερωτικέ στήλες με πληροφορίες για τις τιμές, ε, τι, τους, τους χρόνους αφήξεων αναχωρήσεων των ε, τρένων. Ε, λίγο πριν από την απόφαση του ρυθμιστικού φορέα λύθηκε και αυτό, μας εδόθησαν. Επίσης υπάρχουν συμβάσεις με κάποιες διαφημιστικές εταιρείες που υπήρχαν συμβάσεις που απαγόρευαν ε, στην Westbahn να κάνει διαφημίσεις ε, και αυτό λύθηκε και άλλαξαν οι συμβάσεις αυτές προς τη δική μας κατεύθυνση. Ε, επίσης, πληροφορίες για χρόνους αφήξεων αναχωρήσεων αυτό το κάλυπτε, η, το μια αυστριακή σιδηρόδρομη για όλους. Εμείς πήγαμε στο δικαστήριο κατά τον, για τα καρτέλ και ολοκληρώθηκε, συμπεριελήφθη και το ε, πρόγραμμα της Westban. Ε, τα, ε, επίσης υπάρχει link για τα εισιτήρια. Ε, αυτό το πρόβλημα με το link εισιτήριο δεν έχει ακόμα επιληθεί. Επίσης ε, θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας τις παλαιές συμβάσεις που ισχύουν και δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος των νέων εισερχομένων. Ε, γιατί πολλές φορές ε, επί τέσσερα χρόνια υφίσταται περιοριστικές διατάξεις. Ε, αυτό το αντιμετωπίσαμε γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να μπαίνει κάποιος νέος στην αγορά. Νομίζω ότι με την σύνοψη που θα κάνω είμαι στο, μέσα στο δεκάλεπτο. Τώρα, προσδοκίες απέναντι στην πραγματικότητα. Ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να προχωρήσουμε, είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά πρέπει να γίνουν πιο πολλά για να μειωθούν οι διακρίσεις. Είναι πολύ σημαντική η υποστήριξη από τον ρυθμιστικό φορέα. Ε, υπολογίζουμε σε αυτόν και είχαμε αποτέλεσμα. Επίσης, χρειαζόμαστε οι ιδιώτες επενδυτές να έχουν με συνθήκες διότι οι απρόβλεπτες ε, εξελίξεις και αυξήσεις του κόστους της υποδομής ε, αλλάζει τα επιχειρηματικά προγράμματα ε, και αυτό είναι καταστροφικό και επίσης θέλουμε πάντοτε να λειτουργούμε με τρόπο φιλικό προς τον πελάτη και δίκαιο απέναντι στον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φώστα. Θα έπρεπε να έχω κάτι να, να σας ειδοποιώ από την οπτική τώρα των ε, κατεστημένων φορέων, ο κύριος Μορέτη, διευθυντής, διοικητής, ε, γενικός διευθυντής του ΕΦΕΣ. Κύριε Μορέτη, 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να σας παρουσιάσω με δύο λόγια τι είναι η οργάνωσή μας, το CR εκπροσωπεί περί τα 80 μέλη, εκ των οποίων 23% είναι ιδιώτες. Το 90% των ε, φορέων, των επιχειρήσεων, για επιβατικές μεταφορές και το 75% και το προγραμμίζω αυτό των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τα δίκτυα. Το λέω αυτό διότι η εσωτερική συζήτηση μας ήταν σύνθετη, διεξοδική και μακρά. Κατέληξε ωστόσο σε κοινά συμπεράσματα μεταξύ τόσο διαφορετικών φορέων με τόσο διαφορετικά συμφέροντα. Η πρόταση που υποβάλλουμε, κοινή πρόταση επαναλαμβάνω στο σενάριο αυτό, δείχνει μια μεγάλη εμπιστοσύνη και μια βούληση να ξεκινήσει ταχύτατα, να υλοποιηθεί ταχύτατα και να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα μπρος σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν μακρά και πολύ διαφοροποιημένη. Υπήρξαν πολλές αλλαγές στον κλάδο ενώ θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν λίγες αλλαγές, καλά φτιαγμένες, με καλή μελέτη που θα δώσει στον κλάδο σταθερότητα, τόσο ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν μια σαφή στρατηγική και να επενδύσουν με βεβαιότητα. Χωρίς αυτό υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχει σωστή, να μην κάνουμε σωστή δουλειά. Οι μεταρρυθμίσεις που υποβάλλουμε έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα, δηλαδή επέτρεψαν στους incumbent ε, μια μεγάλη εξέλιξη. Βλέπετε στον πίνακα την τελευταία επταετία του δικού μου ομίλου που βελτίωσε την οικονομική του κατάσταση κατά 2,5 δις. Το ίδιο έκαναν και άλλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους ε, πελάτες μας, πολίτες που χρησιμοποιούν το τρένο και πελάτες που συμβάλλουν με φόρους ε, στην ε, εξυπηρέτηση των υποδομών ή της δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης, είχαμε και μια μεγάλη είσοδο νεοεισερχόμενων. Το 25% τώρα ανήκει σε newcomers. Ωστόσο, και παρά τα αυτά είχαμε μια μεγάλη ανάπτυξη που, αφε, που μείωσε τις ε, ζημίες από τα 18,5% στα 16,5%. Τι δεν λειτουργεί δεν λειτουργεί, το ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τον κλάδο αυτό ως ένα κλάδο απομονωμένο από τους υπόλοιπους. Πρέπει να τον δούμε στο πλαίσιο ε, συνολικά των μεταφορών και να δημιουργηθούν κανόνες ανταγωνισμού διά λειτουργική πιο δίκη, με μεγαλύτερες δυνατότητες του να μπορεί να κάνει κάποιος επιχειρηματική δραστηριότητα με παρόμοιες υποδομές και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Τα τελευταία 20 χρόνια κάναμε πολλούς δρόμους, λίγους δρόμους και αυτό είχε συνέπειες. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε η προσέγγιση μας του σιδεδρόμου να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο πλαίσιο της ε, διατροπικότητας των μεταφορών. Επίσης, είχαμε προσπαθήσει να ανοιχτούμε στους επιβάτες με μικρή επιτυχία. Και γιατί αυτό στους διεθνείς μεταφορές επιβατών. διότι κυρίως δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε στις εμπορευματικές μεταφορές σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλά εμπόδια. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο το χέο υλικό πρέπει να το φτιάξουμε σχεδόν μέτρο-μέτρο. Δεν υπάρχει ένας ε, ανάδοχος που μπορεί να, το, να, να παράσχει ενιαίο τροχαίο υλικό όπως συμβαίνει σε άλλα μέσα μεταφορών όπως τις οδικές. Έχουμε τεχνικά εμπόδια και γραφειοκρατικά εμπόδια. Η διεθνοποίηση της του επιβατικού κοινού δεν προχώρησε κυρίως για, πολλούς ε, γραφειοκρατικούς, για πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια που δεν δέχονται το, τη διέλευση των συνόρων. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το προεξοφλήσουμε στο τέταρτο πακέτο ενδεχόμενα για να μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε τα δύο προβλήματα που ήδη λύσαμε. Εμπορεύματα και επιβάτες λαμβάνοντας υπόψη τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Κάτι ακόμα που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει πριν μπούμε στην ουσία του τέταρτου πακέτου είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Εμείς είμαστε υπέρ της υποστήριξης του ανοίγματο του στους επιβάτες της εθνική, των εθνικών μεταφορών και νομίζω ότι όλος ο κλάδος το συμμερίζεται. Είχαμε μια μεγάλη επαναλαμβάνω εσωτερική συζήτηση η οποία παρουσιάζει μια κοινή θέση που την υποβάλλει στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Το τέταρτο πακέτο πρέπει να έχει και άλλο στόχο. Να δημιουργήσει σταθερότητα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αλλαγέ κάθε δύο χρόνια. Πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα μιας μακράς σύνθετης διαδικασίας που θα πρέπει να δώσει ένα σαφή πλαίσιο, ένα σαφές πλαίσιο για μια μακρά περίοδο, ούτω ώστε ο επιχειρηματίας να αξιολογεί την αγορά και να επενδύσει χωρίς να φοβάται ότι θα ανακύψουν άλλες αλλαγές. Επίσης πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ποιότητα των συνδρομικών υποδομών, όχι μόνο ποσότητα και ποιότητα, ομοιογενούς χαρακτήρες ευρωπαϊκού ευρωπαϊκό υπάρχουν εμπόδια στα σύνορα, να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, ρυθμιστικών αρχών σε εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών αρχών, όπου θα υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής εμπειριών και όπου ιδίω θα μπορούν να γίνουν ομοιογενείς οι εθνικοί κανόνες βάσει των ευρωπαϊκών ενδείξεων που το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να δώσουν, οπωσδήποτε. Σε ό,τι αφορά το πακέτο, το πρώτο πρόβλημα που τέθηκε ήταν της αξιολόγησης της ποιότητας της πρότασης. Της αξιολόγησης δηλαδή κατά βάση του impact assessment που παρουσίασε η Επιτροπή ε, στην πρότασή της για το τέταρτο πακέτο. Δεν το κάναμε μόνοι μας, το κάναμε τη βοήθεια γνωστών ε, επαγγελματιών του χώρου που είναι ανεξάρτητοι και φημισμένοι για την εξάρτησή τους μεταξύ του Imperial College και το TAFT, το Πανεπιστήμιο TAFT που συνθετικά μας είπαν ότι η πρόταση δεν είναι μια δυνατή πρόταση, δεν είναι μια πρόταση που βασίζεται σε σαφή γεγονότα, σαφή αποδεκτικά στοιχεία, δεν είναι πρόταση που λαμβάνει υπόψη την επιστημονική έρευνα και συζήτηση που έγινε μετά από εμπειρία που διαπιστώθηκε επί τόπου. Είναι μια πρόταση που επιλέγει κάποια παραδείγματα για να μπορέσει να καταλήξει στο να αυτοαναδεικνύει τον αρχικό της στόχο που είναι κάπως ε, πρόκριμα ε, αυθαίρετο πρόκριμα αν δεν στηρίζεται σε αποδεκτηρευμένα στοιχεία. Παράδειγμα είναι το θέμα της αύξησης της εκμετάλλευσης των δικτύων. Τούτο, αυτό ήταν το βασικό εργαλείο, ο βασικός στόχος της πρότασης, αλλά έγινε μόνο μιλώντας για τον κλάδο των επιβατών. Στα ίδια, στις ίδιες γραμμές ωστόσο περνάνε και τα εμπορεύματα. Περνάς λοιπόν από, την υψηλή, από το υψηλό αριθμό που δίνει η Επιτροπή για τους επιβάτες στο χαμηλό αριθμό για τα, εμπο, για τα εμπορεύματα. Ε, προσθέτω εγώ. Αν αντί κάναμε αντιπαραβολή όχι με χιλιόμετρο αναγραμμή αλλά, αλλά α, χιλιόμετρα ανά ε, γραμμή τρένου θα είχαμε διαφορετικά στοιχεία. Στην Ιταλία υπάρχουν 16.000 ε, γραμμές, 16.000 χιλιόμετρα γραμμής, αλλά είναι διπλή γραμμή, άρα διπλασιάζουμε τον αριθμό. Αν αλλάξει λοιπόν τον τρόπο υπολογισμού, αλλάζει και τα αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν ε, ζητούμε να επανεξεταστεί η βάση υπολογισμού των προτάσεων, αλλά και το σκεπτικό των προτάσεων της Επιτροπής. Οι δικές μας προτάσεις ποιες είναι. Ας πούμε σε πιο σύνθετα θέματα. Το unbundling, ο διαχωρισμός. Ε, η προσέγγιση της Επιτροπής μας φαίνεται υπερβολικά δογματική, κυρίως όμως που δεν βασίζεται σε μια αποδεδειγμένη, ισχυρή βάση. Εμείς προσπαθήσαμε να στηριχθούμε εδώ σε μια σειρά σημαντικών ακαδημαϊκών από το Πανεπιστήμιο του Leeds, του Delft, του Κόμπε και παρουσιάσαμε μια μελέτη που είναι στη διάθεσή σας. Προσπαθήσαμε να δούμε στην πράξη την οικονομική βιωσιμότητα της πρότασης αυτής. Η απόδειξη είναι ότι με την υφιστάμενη πυκνότητα του ευρωπαϊκού δικτύου θα υπήρχε αύξηση κόστους κατά 6 δις. Και το ερώτημά μας είναι ποιος θα πληρώσει. Πριν μπούμε στην ουσία, αυτά τα 6 δις θα φορτωθούν το εισιτήριο των επιβατών, τους τόνους ε, ε, ε, εμπορεύματος, το φορολογούμενο. Πώς υποστηρίζεται η αύξηση αυτή. Αν ακολουθήσουμε κατόπιν το ευκταίο για μας στόχο της Επιτροπής να αυξηθεί η συχνότητα εκμετάλλευση, πυκνότητα εκμετάλλευσης του δικτύου, σύμφωνα με τους στόχους της Επιτροπής, η αύξηση του κόστους του unbundling θα έφτανε τα 15 δις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τεράστια νούμερα που πρέπει να αιτιολογηθούν για να αποφύγουμε πριν φτάσουμε σε απόφαση να υπάρχουν λύσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε το πρόβλημα των νέων εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών. Να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τα δίκτυα εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα διασυνοριακά, και να βρούμε έναν τρόπο που θα επιτρέπει κάθε μορφή λύσης ουσίας να ανατίθεται στα κράτη-μέλη και να οδηγεί βάσει σαφών ενδείξεων που θα πρέπει να δώσει η Επιτροπή Κοινοβούλιο σε μια ισότιμη, ισοδύναμη ανάλυση της οικονομικής βιώσιμότητας των λύσεων που θα επιλεγούν. Μπορείτε να κλείσετε, λέει ο Πρόεδρος, αμέσως. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση της πρόσβασης ε, στο εθνικό επιβατικό δίκτυο είμαστε υπέρ, αλλά αυτό θα πρέπει να εξισορροπηθεί με την ισορροπία της παροχής δημόσιας υπηρεσίας, που είναι φυσικό. Αλλιώς θα υπήρχαν εμπόδια Αμφισβήτηση της ελεύθερης πρόσβασης. Είναι λοιπόν προς όφελος όλων να βρεθεί μια στέρεη λύση στο σημείο αυτό. Προσθέτουμε ωστόσο ότι στη μεταβατική περίοδο, γιατί ξεκινάμε από διαφορετικές εμπειρίες, θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος αμοιβαιότητα στην ε, δραστηριοποίηση, μεταβατική σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, αλλά μόνιμο μεταξύ επιχειρήσεων που έρχονται από έξω ευρωπαϊκές χώρες, γιατί ήταν παράλογο να ανοίξουμε εμείς ε, το, την αγορά μας χωρίς να ζητήσουμε αμοιβαιότητα. Να κλείσω με τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματά μας είναι η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά με μια σειρά στέρεων οικονομικών δεδομένων, ιδίως στην οικονομική βάση, και να γίνει επιλογή που πηγαίνει προς τη δημιουργία μια ενιαία αγορά το συντομότερο δυνατό με αμοιβαιότητα σε μεταβατικό επίπεδο, αφήνοντας τα κρατη το πρόβλημα του unbundling, υποχρεωνώντας ωστόσο να έχουν πλήρη διαφάνεια και ενισχύοντας τις ρυθμιστικές αρχές για να υπάρχει βεβαιότητα σε όσους θέλουν να μπουν στην αγορά. Κρίνω ο συνάδελφος είναι σε ένα κράτο όπου υπάρχει μια ενοποιημένη επιχείρηση. στι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη, ωστόσο, η δραστηριοποίηση γίνεται στην Γερμανία και την Ιταλία. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα όπου υπάρχει ανταγωνισμό στο, στην υψηλή ταχύτητα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει απελευθέρωση και υπό του όρου αυτού, Μπορεί να γίνει, ωστόσο, και με σεβασμό τη οικονομική βιωσιμότητα που είναι βασικός, βασική προπόθεση τη επιχειρήση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Μωρέτη. Βλέπω ότι θα είναι δύσκολη η δουλειά του Προέδρου γιατί δεν περιορίζεστε στο δεκάλεπτο. Σας ξαναπαρακαλώ να σέβεστε το χρόνο που σας δόθηκε. Επόμενος. Τα εμπορεύματα. Έχουμε τον πρόεδρο του Rail Freight της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις συνθήκες ανάπτυξης των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων και τα επιπτώσεις της σχετικής δέσμης μέτρων. Δεν θα μιλήσω για το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί τα λέμε αυτά στην ιστοσελίδα μας, καθώς ε, όπου θα βρείτε και τα έγγραφα της σημερινής ακρόασής μου η μεταφορά εμπορευμάτων από τους σιδηροδρόμους στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε 7 επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Ποιες είναι λοιπόν οι συνθήκες για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Είναι κάτι πολύ απλό. Η κυκλοφορία των εμπορευμάτων έχει απελευθερωθεί όπως ξέρετε και νομίζω ότι πρέπει να έχει τις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού με τους υπόλοιπους τομείς για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις οδικές μεταφορές. Πρόκειται λοιπόν για μια ενιαία αγορά μέσα στην οποία να μπορέσουν οι σιδηρόδρομοι να είναι ανταγωνιστικοί. Θα έπρεπε να υπάρξει ένα ενιαίο είδος σιδηρογραμμής. Θέλουμε λοιπόν μια ενιαία αγορά και για τους σιδηροδρόμους. Και αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι πρέπει να υπάρξουν αρκετές επιχειρήσεις για να υπάρχει ανταγωνισμός. Δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και γι' αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι λιγότερο το αρχικό κόστος για τους χρηματοδότες και τους μετόχους να έχουν δηλαδή επαρκή έσοδα και την βεβαίωση ότι δεν θα βλαφτούν τα συμφέροντά τους ξαφνικά λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας ή των ε, μέτρων. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι χρειάζεται μία διαχείριση των υποδομών με συνεπή πολιτική και συγκεκριμένες και σαφείς ευθύνες, δίκαια πρόσβαση στο σύστημα και δίκαια και λογικά ναύλα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη συνεργασίας των διαχειριστών των επιχειρήσεων αυτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και τέλος πρέπει να υπάρχει συνδυασμός των συστημάτων μεταφορικών ικανοτήτων κλπ. Κοινά δηλαδή ευρωπαϊκά πρότυπα που τα εφαρμόζει και τα καθορίζει η ΕΡΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων, που χρησιμοποιούν φυσικά υπεργολάβους. Βέβαια το κυριότερο κριτήριο είναι ο δίκαιος ανταγωνισμός και πρέπει να υπάρχει και μία αρχή στην οποία να προσφεύγει κανείς. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Μωρέτη, δεν χρειάζονται περισσότερες μελέτες ούτε για το κόστος ούτε για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται μία ενιαία αγορά λειτουργική για τους σιδηροδρόμους. Τώρα για τη δέσμη των σιδηροδρομικών μέτρων. Θα την περιγράψω με όρους governance. Πρέπει να υπάρχει πλήρης λογοδοσία, καθορισμός διαφανής των ωραρίων κλπ και σωστός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ μετόχων και πελατών και σωστός συντονισμός βέβαια και από την Κομισιόν και τις κυβερνήσεις. Για να δημιουργηθούν σωστές συνθήκες ανταγωνισμού, δίκες, εμείς δεχόμαστε τον πλήρη διαχωρισμό που προτείνεται να μην υπάρχουν ειδικέ προτεραιότητες για τα ωράρια και την πρόσβαση. Ας μην επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις υποφέρουν πολλές φορές από τέτοια μέτρα. Ούτε χρειαζόμαστε κρυμμένες επιχορηγήσεις. Θεωρούμε ότι χρειάζεται διαχωρισμός του προσωπικού των γραφείων και των επιχειρήσεων που ήδη υπάρχουν γιατί αυτό είναι ένας σωστός τρόπος να αρχίσουμε τα πράγματα. Ίσως να μην χρειάζεται να εφαρμοστεί και μακροπρόθεσμα, αλλά είναι μια αρχή. Πριν από ένα χρόνο, ακούσατε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι πρέπει να υπάρξει ο πλήρης διαχωρισμός και μόνο μετά θα μπορούσε να αρχίσει η συνεργασία. Φυσικά χρειάζονται και ανεξάρτητα, ανεξάρτητες οργανώσεις και υπηρεσίες εποπτείας. Δεν δεχόμαστε τη συνέχιση του υπάρχοντος προτύπου γιατί νομίζουμε ότι αυτό θα πνίξει τον ανταγωνισμό. Και τουλάχιστον πρέπει να υπάρξουν ορισμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεών του αλλά οι προτάσεις της Κομισιόν ως έχουν χρειάζονται περισσότερη ενδυνάμωση. Γιατί αυτή τη στιγμή ένα κράτος μέλος μπορεί να προσφύγει λέγοντας ότι δεν δέχεται την πρόσβαση της Α ή της Β επιχείρησης στο, στην επικράτειά του, των τρένων της επιχείρησης. γιατί οι ανεξάρτητες υδρονομικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν νομίζουμε την ε, δυνατότητα να προσφεύγουν και στην Κομισιόν, όχι μόνο η μία χώρα στην άλλη. Δεν είναι ο σωστός τρόπος αυτός. Είναι λοιπόν μια σοβαρή πρόσθετη ρήτρα εδώ που απαιτείται αν θέλουμε να επιβιώσει το πρότυπο. Τέλος, ξέρω ότι θα τα πείτε και το απόγευμα, αλλά πρέπει η ενιαία αγορά για να λειτουργήσει να έχει πλήρη δια... να υπάρχει πλήρη διασύνδεση των συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη με έναν ενιαίο, με ενιαίους κανόνες και πρότυπα που πρέπει να τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων με τις εθνικές αρχές ασφαλείας, οι οποίες όμως θα είναι σαν υπεργολάβοι όπως είπα και προηγουμένως, για να διασφαλίζουν απλώς την σωστή μεταφορά των προτύπων από χώρα σε χώρα. Όχι όμως και εθνικά πρότυπα, ενωσιακά μόνο. Εκτός αν είναι κάτι τελείως απαραίτητο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ξέρετε, έχουμε μικρότερο εύρος των γραμμών. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Οι επιχειρήσεις όμως δεν ε, ανησυχούν από αυτό, λένε θα κάνουμε και μικρότερα βαγόνια. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ε, ενιαία πρότυπα που να τα καθορίζει η Ευρωπαϊκή αυτή αρχή συντηροδρόμων και ένα καλό συμπέρασμα είναι η ατμομηχανή της τάξεως 96. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι για να καταλήξω θα έλεγα ότι υποστηρίζω την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους γιατί νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να ανοίξει την αγορά και τα δίκτυα στον ανταγωνισμό. Έτσι θα υπάρξουν νέες ιδέες, νέες αποτελεσματικότητες, ιδιωτική επένδυση και άρα ανάπτυξη. Αυτά τα χρειαζόμαστε όλα, αλλά πρέπει οι επενδυτές να έχουν τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν καταχρήσεις ή δεν θα ζημιωθούν από νομικούς φραγμούς που θα τεθούν αυθαίρετα από κράτη για τα, να προστατέψουν τα συμφέροντά τους. Χρειάζεται δίκαιος ανταγωνισμός, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε μερικές χώρες μέλη και γι' αυτό σε αυτές δεν υπάρχουν τόσο, πολύ ανεξάρ, τόσο πολλές ανεξάρτητες ιδρυνομικές επιχειρήσεις. Βέβαια υπάρχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, αλλά πώς γίνεται να αγοράζονται μικρότερες εταιρείες από Πού τα βρίσκουν τα λεφτά σε αυτά τα κράτη τουλάχιστον. Καταλήγω λοιπόν λέγοντας ότι είναι ουσιώδες για μας τα μέτρα της τέταρτης δέσμης να εφαρμοστούν ως σύνολο, χωρίς αποδυνάμωση, με ενθάρρυνση του δίκαιου ανταγωνισμού και άρα οι αλλαγές πρέπει να γίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη με πλήρη διαφάνεια και λογικό χρονοδιάγραμμα. Έτσι μόνο θα υπάρξει η σταθερότητα για την οποία μίλησε προηγουμένως ο κύριος Μωρέτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Τόνι. Τώρα, ακολουθεί η προοπτική του διαχειριστή των υποδομών. Η Μόνικα Χάιμινγκ θα μας μιλήσει, είναι εκτελεστική διευθύντρια της EIM ε που είναι οι Ευρωπαίοι διαχειριστές σιδηροδρομικών υποδομών. Ευχαριστώ πολύ, Μπράιν. Όχι, δεν έχω διαφάνειες. Κάποια σημαντικά σχόλια θέλω να κάνω. Οι διαχειριστές χαίρομαι που έχουν φωνή εδώ. Είμαστε ευτυχείς για την πρόσκληση. Τα μέλη της EIM πιστεύουν στην πρόταση, ε, την τέταρτη δέσμη μέτρων, που είναι αποτέλεσμα αναγκών που εντοπίστηκαν νωρίτερα στην αγορά. Κάποιοι μπορεί να πείτε, α, πολύ ωραία έχουμε το την πρώτη δέσμη, τη δεύτερη, την αναδιατύπωση. Γιατί να έχουμε και τέταρτη δέσμη μέτρων. Η τέταρτη δέσμη μέτρων γεμίζει τα κενά που υπήρχαν και γι' αυτό ε, ο CIM είμαστε σαφώς υπέρ της τέταρτης δέσμης και επειδή είμαστε και στο πίεσο που δεν είναι το δικό μας θέμα, ε, τα αφήνουμε στους, διαχει... στους επιχειρηματίες, ε, στις επιχειρήσεις. Το κομμάτι της διακυβέρνησης μας απασχολεί εμάς πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό. Η συζήτηση πάνω στη διακυβέρνηση θα πρέπει να εστιάσει στον ρόλο των διαχειριστών στο μελλοντικό σύστημα μεταφορών. Ο ρόλος του διαχειριστή υποδομών είναι συστημικός ρόλος δεν μπορούμε λοιπόν να ε, περιοριστούμε σε ένα κομμάτι, γιατί όταν δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχουν σειρμοί, δεν υπάρχει ε, τοπική μεταφορά. Ε, είναι η αρχή και το τέλος. Και στη Γαλλία ακόμα έχουμε μεγάλη μεταρρύθμιση στους σιδηροδρόμους που δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί, αλλά ένα στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και εκεί και μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος ε, είναι η ένταξη και ο συντονισμός των διαχειριστών υποδομών. Γι' αυτό είναι σοφή απόφαση και τη στηρίζουμε. Η πρόταση της Κομισιόν ε, βάζει έμφαση στο πώς θα πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοση των διαχειριστών υποδομών. Και αυτό θέλουμε να γίνει και θέλουμε να ε, δώσουμε έμφαση εκεί. Τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας, όπως είπατε κι εσείς. Έχουμε τους χρήστες, έχουμε τις περιφέρειες, έχουμε τους πολίτες. Και εμείς ως διαχειριστές υποδομών λέμε, ωραία, η πρόταση για τη διακυβέρνηση της Κομισιόν περιλαμβάνει κάποια κρίσιμα στοιχεία που, για να ε, ανταποκριθούμε στις αποδόσεις που αναμένονται από εμά και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και θα πρέπει να δουλέψουμε με τρόπο μετρήσιμο, διαφανή και όλοι θα πρέπει να κάνουμε σχόλια. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης. Αυτά είναι πράγματα που μας βρίσκουν σύμφωνους ως EIM και ως μέλη και τα μέλη της EIM συμφωνούν για τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, που είναι κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ποιοτικού δείκτες. Οι ποιοτικοί δείκτες είναι πολύ σημαντικοί για την μεγαλύτερη απόδοση, πρέπει να είναι διαφανείς και μετρήσιμοι. Οπότε, ε, Εμεί ε, δεσμευόμαστε απόλυτα να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά ως EIM γιατί θα δώσει ωφέλη και για το σύστημα και για τους πελάτες και για τους ιδιοκτήτες και για τις περιφέρειες και πιστεύουμε ότι τα θέματα αυτά για την απόδοση και το πώς θα ε, επιτύχουμε την απόδοση και πώς θα έχουμε συντηρητική αξιολόγηση, όλα αυτά θα καθορίσουν το ρόλο των σιδηροδρόμων στο μέλλον και θα επηρεάσουν και την πολιτική μετα... σιδηροδρομικών μεταφορών. Και πάμε ακόμα παραπέρα ως ε, ανεξάρτητοι διαχειριστές ε, ε, αποδεικνύουμε ότι γίνεται να είναι ανεξάρτητοι διαχειριστές υποδον μπορούν να έχουν καλές επιδόσεις. Εμείς είμαστε η απόδειξη ζωντανή ότι η ανεξαρτησία έχει αποτέλεσμα. Καταλαβαίνουμε και την ανάγκη να συνεργαστούν οι διάφοροι δραστηριοποιούμενοι στον κλάδο εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, να είμαστε φιλικοί προς τον χρήστη, προς τους χρήστες με διαφανή και ανοιχτό τρόπο. Θα πρέπει να έχουμε ε, σαφή ρόλο, ε, σαφείς αρμοδιότητες και λειτουργίες ε, για να συνεργαζόμεθα στενότερα με ξεκάθαρο τρόπο και χωρίς διακρίσεις. Πιστεύουμε ότι οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται ε, ισότιμα σε όλη την Ευρώπη, ε, όχι εμπαλωματικά. Γι' αυτό χρειάζεται η τέταρτη δέσμη μέτρων για να λυθούν αυτά. Δεν πρέπει να έχουμε δύο παράλληλα καθεστώτα είτε ε, υπάρχει είτε δεν υπάρχει ολοκληρωμένος διαχείριση συστημάτων. Πρέπει να έχουμε ε, μία δέσμη μέτρων που θα γίνονται κατανοητά με τον ίδιο τρόπο και θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο παντού. Γιατί το χειρότερο είναι αυτή η εμβαλωματική προσέγγιση στην Ευρώπη με διαφορετικές ταχύτητες. Αυτά τα παράλληλα καθεστώτα θα πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσμα της τέταρτης δέσμης μέτρων. Δεν πρέπει να έχουμε διαφορετικό τεχνικό μέρος ε, ή διαφορετικές ε, υποδομές. Θα πρέπει να είναι όλα ενιαία. Η συνεργασία είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να υπάρχουν και δια... για να έχουμε και διασυνοριακές υπηρεσίες που θα παρέχονται με τον ίδιο τρόπο ε, θα αξιολογούνται συγκριτικά με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε απρόσκοπτη ενιαία Ευρώπη, ομαλή, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομών. Αλλιώς δεν γίνεται. Και η πρόκληση για τον κλάδο είναι να αποδείξει ότι ε, είναι ικανός να τα ε, παραδώσει όλα αυτά. Εμείς χαιρόμαστε που μπορούμε να το κάνουμε και υπάρχουν και συνεργασίες μεταξύ ρυθμιστικών φορέων και άλλων εμπλεκομένων. Ή Οι και περιφέρειες να συνεργάζονται στην ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών, στη συγκριτική αξιολόγηση και εμείς μπορούμε να το κάνουμε ως ε, διαχειριστές υποδομών. Και τέλος, πολύ σημαντικό, μια και είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μήνυμα προς τους ε, ευρωβουλευτές. μην χωρίσετε το, τη δέσμη μέτρων. Όλα τα στοιχεία στο, στην τέταρτη δέσμη μέτρων είναι αλληλένδετα δεν μπορείτε να ε, ε, κάνετε επιλογή. Γιατί μέτρων, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όλα τα τμήματα είναι λιλένδετα και αφού όλα τα τμήματα τα δείτε, όλα τα μέρη της δέσμης, θα καταλήξετε σε μια αξιοπρεπή πρόταση που θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με τρόπο ασφαλή για την αγορά, ούτως ώστε να αποδειχθεί λειτουργική και να έχει αποτέλεσμα. Μην βγάλετε ένα τμήμα, ε, προχωρήστε με βάση ολόκληρο το πακέτο. Εμείς το χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε τη δέσμη αυτή γιατί όπως είπα συμπληρώνει τα κενά που λείπουν, τα κλείνει και βέβαια αν δεν γίνει σωστά η δουλειά θα υπάρξει και πέμπτη και έκτη και έβδομη δέσμη μέτρων. Αυτό δεν θα ήταν καλό. Δεν μπορούμε μια ζωή να ασχολούμεθα με, τα, με τις δέσμες μέτρων. Θα, το, θα ασχοληθούμε μια φορά για να γίνει σωστά η δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Μόνικα, όλοι ελπίζουμε να μην υπάρχει πέμπτη, έκτη, έβδομη δέσμη. Γιατί... Ε, θα πρέπει βέβαια να καλύψω ε, καλύψουμε τα νότα μας, ε, ούτως ώστε να αποφύγουμε να ασχολείται και η 15 μηνών εγγονή μου μετά την ένατη δέσμη, δέσμη μέτρων. Η Ζαμπίνε Τριέρ είναι η επόμενη ομιλήτρια που θα μας παρουσιάσει την προοπτική των εργαζομένων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι παρακολουθώ την τέταρτη δέσμη και έχω ήδη κουραστεί από την τέταρτη δέσμη. Εγώ νομίζω ότι δεν μας χρειάζεται. Το ETF εκπροσωπεί 150.000 ε, εργαζόμενους ε, όλων των επαγγελμάτων στον τομέα. Και η αρχική μου παρατήρηση είναι ότι τελικά όταν μιλούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφαλή λειτουργία των σειροδομικών υπηρεσιών χρειαζόμαστε προσωπικό με εμπειρία, ικανότητες, σωστές συνθήκες εργασίας ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν σωστά και με ασφαλή τρόπο τη δουλειά τους και προσωπικό που έχει κίνητο να δουλέψει. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσετε όταν αποφασίζετε για το νομοθετικό πλαίσιο. Ξεκινώ τώρα με την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας. Η βάση, την πρόταση αυτή. Το βασικό στοιχείο της πρότασης είναι να επιβάλλει ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς για όλες τις επιβατικές υπηρεσίες στην Ευρώπη ως την μόνη υφιστάμενη επιλογή και να καταργήσει για τον σειροδομικό τομέα την υφιστάμενη δυνατότητα των κρατών και των αρμόδιων αρχών να επιλέγουν μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων είτε διαγωνισμό είτε απευθείας ανάθεση. Θέλω να σας θυμίσω ότι για να περάσει ο κανονισμός αυτός χρειάστηκαν 7 χρόνια και τρεις διαφορετικές προτάσεις της Επιτροπής. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήδη προσπάθησε να επιβάλλει ανταγωνιστικό διαγωνισμό ως την μόνη επιλογή που απορρίφθηκε στην φάση της νομοθετικής διαπραγμάτευσης. Ο υφιστάμενος κανονισμός υιοθετήθηκε τέθηκε σε ισχύ το 2009 μόνο και βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο τμήμα, στο πρώτο ήμιση της μεταβατικής περίοδου που λήγει το 2019. Τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν μια ενδιάμεση έκθεση το 2014-2015 και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει ακόμα αρχίσει να λειτουργεί. Γιατί να το αλλάξουμε. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η επιβολή ενιαίας και μίας δυνατότητας για την οργάνωση των συνδρομικών υπηρεσιών είναι, υπηρεσιών είναι κατά του, άρθρου, του πνεύματος του άρθρου 14 και του πρωτοκόλλου 26 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που αναφέρεται, όπου αναφέρεται σαφώς ότι τα κράτη-μέλη και οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα επιλογής για να αποφασίσουν το πώς θέλουν να οργανώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους. Η επιλογή για το πώς θα οργανωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες σημαίνει ότι είτε αυτό θα γίνει με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο του υφιστάμενου κανονισμού ή μέσω ανταγωνιστικού διαγωνισμού. Κατά την άποψή μας λοιπόν αυτό αντίκειται στο πνεύμα των άρθρων αυτών και του πρωτοκόλου 26 να επιβάλλεται μία και μόνο επιλογή. Γι' αυτό η Ομοσπονδία μας ζητά από τα μέλη του Κοινοβουλίου να απορρίψουν την πρόταση του κανονισμού. Επίσης, να τονίσω στο πλαίσιο αυτό το θέμα, το θέμα της κοινωνικής διάστασης που έχει σημασία για τους εργαζόμενους μας που επιτρέπουν να τώρα το να είτε έχουμε ανοιχτή τον ανταγωνισμό με σύμβαση ή με διαγωνισμό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός γίνεται πάντα στο επίπεδο της χαμηλότερης, ε, του χαμηλότερου τιμήματος που σημαίνει για μας ότι μειώνονται οι συνθήκες, ε, οι, οι, συνθήκες εργασίας. Και και η μείωση συνήθως αφορά το μείωση του κόστους του προσωπικού. Στον κλάδο ένα μεγάλο τμήμα του κόστους είναι σταθερό κόστος που δεν μπορεί να αυξομοιωθεί. Το κόστος προσωπικού ωστόσο είναι αυτό που μπορεί να μεταβληθεί ευκολότερα. Για το λόγο αυτό ήδη τώρα διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα περικοπών οδηγούν σε outsourcing που σημαίνει ότι οι, οι δουλειές καλής ποιότητας στο συνδημικό τομέα θα μειωθούν και θα υποστούν πιέσεις οι εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων, ενώ σε πολλά άλλα σημεία η ασφάλεια της απασχόλησης τίθεται επαμφιβόλο, οι εργαζόμενοι ζουν σε ανασφάλεια όταν αναγγέλλονται οι διαγωνισμοί, δεν ξέρουν δηλαδή αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν ή όχι. Υπάρχουν λοιπόν αρνητικές, πολλές αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους. Στον υφιστάμενο κανονισμό υπάρχει, υπάρχουν ήδη άνθρωποι που δίνουν την ευκαιρία να μειωθούν οι επιπτώσεις αυτές. Το άρθρο 4.5 και 4 6 μιλούν για την προστασία του προσωπικού σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών διαγωνισμών και την δυνατότητα επιβολής ποιοτικών κριτηρίων που περιλαμβάνουν και εργασιακά και κοινωνικά κριτήρια. Το πρόβλημά μας είναι ότι το άρθρο αυτό δίνει στην αρμόδια αρχή μόνο μία επιλογή για να δεν αποτελεί υποχρεωτικό κανόνα. Αφετέρου επειδή ο στόχος είναι η μείωση του κόστους, μπορεί να φανταστεί κάποιος πόσες ε, αρχές ε, χρησιμοποιούν, αν αρχές χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή. Κατά την άποψή μας λοιπόν, όταν υπάρχει ανταγωνιστικός διαγωνισμός και η εργασιακή προστασία του προσωπικού πρέπει να γίνει υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει και, στα δύο, και στις δύο φάσεις του διαγωνισμού, όταν καταγράφονται όταν δημοσιεύονται οι όροι του διαγωνισμού και αφετέρου όταν υπάρξει πραγματικά αλλαγή του ε, φορέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει προστασία του προσωπικού. Για μας είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στο προσωπικό μας πώς είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ευρωπαϊκά όργανα, οι ευρωπαίοι νομοθέτες να επιβάλλουν τον ανταγωνισμό να επιβάλλουν τον κατακαιρματισμό του κλάδου, την αναδιάρθρωσή του αφενός, αλλά από την άλλη όταν μιλούν για την προστασία του προσωπικού να λένε «Α, αυτό δεν είναι θέμα δικό μας, είναι επικουρικότητα». Οι, οι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν τις διαφορές αυτές. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Όταν μιλούμε για την ε, οδηγία απελευθέρωσης ανοιχτής πρόσβασης, στην άλλη οδηγία, στην ανδιατυπωμένη οδηγία μιλώ, αυτό σημαίνει για μας ότι επιτρέπεται να επιλέγει ο καθένας ό,τι καλύτερο θέλει. Ο ανταγωνισμός προφανώς γίνεται μόνο με γραμμή με βάση το κέρδος, μόνο την κερδοφορία. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι όταν υπάρχει, αν λάβετε υπόψη ένα σιδηροδρομικό σύστημα που είναι δίκτυο, που πρέπει να λειτουργεί ως δίκτυο για να παρέχει υπηρεσίε ποιότητα στον επιβάτη και να πηγαίνει και στην πιο απόμακρη περιοχή ή στην πιο μικρή πόλη, χρειάζεται να δούμε το σύστημα ως δίκτυο. Ο ανταγωνισμός ανοιχτής πρόσβασης δίνει την επιλογή ε, της πιο προσοδοφόρας γραμμής χωρίς την σύνδεση ε, με λιγότερο απροσοδοφόρες ε, γραμμές με αποτέλεσμα στις λιγότερο ελκυστικές γραμμές να μην υπάρχει προσφορά. Εάν οι αρχές πούν ότι χρειαζόμαστε τις γραμμές αυτές, τότε πρέπει να το πληρώσουν. Τι γίνεται στην πραγματικότητα, ε, οι προσοδοφόρες γραμμές πηγαίνουν στους ιδιώτες και το δημόσιο φορολογούμενος πληρώνει για τις υπόλοιπες. Επίσης, να σας πω κάτι για το θέμα της διακυβέρνησης. Η οργάνωσή μου είμαστε κατά της του πλήρους διαχωρισμού υποδομών και λειτουργία. Είμαστε υπέρ των ενοποιημένων εταιριών και είμαστε και δεν θεωρούμε ότι η δεύτερη επιλογή αυτή του κινέζικου τείχους είναι χρήσιμη διότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τις ε, συνέργειες ενός ενοποιημένου συστήματος. Υποστηρίζουμε τα επιχειρήματα που λένε ότι δεν υπάρχει εμπειρική εμπειρική απόδειξη ότι ο διαχωρισμός είναι καλύτερη επιλογή αυτή καθε αυτή. Υπάρχουν περισσότερες δαπάνες, μεγαλύτερη κίνδυνη και οι συνέργειες ενός ενοποιημένου συστήματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, να παρουσιάσω την άποψη και την ενσυχία των ε, συνδικάτων ο πλήρης διαχωρισμός θα καταστρέψει την εσωτερική αγορά εργασία μέσα στους ομίλους που είναι ουσιαστικού χαρακτήρα για να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της αναδιάθρωσης. Οι σιδηροδρομικοί υποφέρουν ανά την Ευρώπη από την αναδιάθρωση εδώ και 20 χρόνια. Σε κάποιες χώρες περισσότερα χρόνια, σε κάποιες χώρες το βιώνουν λιγότερα χρόνια, αλλά συνολικά όλοι οι ισοδομικοί υφίστανται μόνιμη αναδιάρθρωση εδώ και 20 χρόνια. Και αυτό είναι κατά βάση αναδιάρθρωση που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όταν λοιπόν η ευρωπαϊκή νομοθεσία καταστρέφει και την εσωτερική αγορά εργασίας, που είναι το μόνο εργαλείο μείωση των, επιπτώ, επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης, πραγματικά αυτό θα είναι κάτι που δεν το καταλάβουν οι σιδηροδρομικοί. Κάτι ακόμα όπου χρειαζόμαστε την εσωτερική αγορά εργασιακή δίνει προοπτική στις ομάδες εργαζομένων που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά του πια, όπως σιδηροδρομικού που έχουν θέματα, που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας και πρέπει να παίρνουν ε, ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις. Συχνά δεν μπορούν να δουλέψουν μέχρι την ηλικία συνταξιοδότηση για ιατρικούς λόγους. Υπάρχει λοιπόν εσωτερική κινητικότητα που τους επιτρέπει ασφάλεια εργασίας. Να τελειώνετε, λέει ο πρόεδρο. Ναι. Μια παρατήρηση. έχουμε να πούμε και για τα θέματα ασφάλειας. Δυστυχώς δεν, έχουμε την, δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε το απόγευμα γιατί θέλαμε και εκεί να πούμε δύο-τρεις παρατηρήσεις. Να έχω δύο λεπτά ακόμα. Όχι. Όχι. Αλλιώς θα συνεχιστούμε, θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ κλείστε. Νομίζω ότι είπα το βασικό μήνυμα. Μην ξεχνάτε την ασφάλεια και το προσωπικό. Για τους ιδεοδόμους αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Χαίρομαι που δεν μιλήσατε μόνο για την ασφάλεια γιατί εδώ ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και είμαι βέβαιος ότι και οι βουλευτές ε, με μεγάλη χαρά θα δέχονταν οποιοδήποτε έγγραφο τους υποβάλλατε σχετικά. Τώρα για τους επιβάτες. Ο Ζαν Πολ Ζακό που είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας των χρηστών των μεταφορικών μέσων. Δέκα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ομοσπονδία μας αντιπροσωπεύει 150 οργανώσεις, 65.000 μέλη συνολικά και ασχολείται με την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών συνεργάζεται με την European Passengers Federation και ασχολείται και με την προστασία του περιβάλλοντος γιατί ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορές και Περιβάλλον. Τρία στοιχεία θα αναφέρω. Πρώτον, ο επιβάτης χρησιμοποιεί δίκτυο που αποτελείται από διάφορους τρόπους μετακίνησης, και χρησιμοποιεί πολλά δρομολόγια. Δεύτερο, χρειάζεται πλήρη και ανεξάρτητη πληροφόρηση και πρέπει να μπορεί να παίρνει το εισιτήριό του από απλά και μοναδικό τρόπο με μονοαπευθυντική θηρίδα. Και τρίτον, έχει απαιτήσει από τις δημόσιες υπηρεσίες για μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Πρώτον, το δίκτυο. Ο επιβάτης χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους μετακίνησης πρώτον τα πόδια του, δεύτερον ποδήλατο, τρίτον το αυτοκίνητό του, σιδηρόδρομο ή αυτοκίνητο. Και όλους αυτούς τους τρόπους πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η επιλογή εξαρτάται από την αρχιτεκτονική των τρόπων αυτών, από την ποιότητα του συνδυασμού των δικτύων, από την ποιότητα των διαφόρων κρίκων της αλυσίδας και από την πληροφόρηση που διαθέτει. Και καταλήγουμε ότι πρέπει να δούμε όλα αυτά τα δίκτυα μαζί. Πρώτον για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του επιβάτη. Δεύτερον για να υπάρχει καλύτερη και μεγαλύτερη κινητικότητα. Ξέρετε ότι υπάρχει γύρανση του πληθυσμού κτλ. Έπειτα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την απαραίτητη μείωση της μόλυνσης και των ε, επιβολών κατά του περιβάλλοντος και τρίτον για να γίνει καλύτερη δυνατή χρήση όλων αυτών των δικτύων δεν περιοριζόμαστε μόνο στους σιδηροδρόμους αλλά στο σύνολο των μέσων μεταφοράς που αλληλοεξαρτώνται. Κάθε σιδηροδρομικό δρομολόγιο πρέπει να εξεταστεί σε σύγκριση με το σύνολο των υπαρχόντων διαφορετικών δικτύων μεταφοράς. και οι κλασικές εταιρείες θα εξεταστούν σε σχέση με το ρόλο που παίζουν σε αυτό το δίκτυο και όχι μόνο ως προς τα συμφέροντά τους. Η πρώτη μας λοιπόν σύσταση είναι να επεξεργαστούμε ένα πολυετές σχέδιο για το σύνολο των μεταφορικών δικτύων με αριθμούς για τις επενδύσεις και τις χρηματοδοτήσεις. Η Νορβηγία, παραδείγματο χάρη, μόλις δημοσίευσε το δεύτερο σχέδιό της για τις μεταφορές, το οποίο θα συντονιστεί ιδιαίτερα, με, θα συνδυαστεί με την προστασία του μη αστικού περιβάλλοντος. Δεύτερη σύστασή μας που προκύπτει από την πρώτη, το σχέδιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από άλλο σχέδιο ειδικά για τους σιδηροδρόμους. από, σε κρατικό βέβαια επίπεδο με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και με σεβασμό των αναλόγων σχεδίων άλλων χωρών. Αυτό το είπαν και πολλοί άλλοι. Ένα συμβούλιο όλων των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα δε των οργανώσεων των επιβατών, θα βοηθάει το κράτος για τη δουλειά αυτή. Και μία ανεξάρτητη οργάνωση θα φροντίζει την επιτήρηση και την εφαρμογή και θα διαχειρίζεται τις πιθανές διαφορές. Δεύτερη πρόταση, πληροφόρηση. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιβατών συνεχώς επιμένει από τότε που υπήρξε η πρώτη οδηγία για τους επιβάτες ότι είναι απαραίτητο οι επιβάτες να έχουν μία και μόνη θηρίδα πληροφόρησης και αγοράς του εισιτηρίου των... Το δεχόμαστε και εμείς. Για να είναι όμως αντικειμενική αυτή η υπηρεσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις επιχειρήσεις. Και αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Οι σταθμοί συνήθως βρίσκονται στα χέρια των εταιριών και πολλές φορές ο επιβάτης πρέπει να πηγαίνει έρχεται σε διάφορα γκισέ για να αγοράσει το εισιτήριό του και αυτό πολλές φορές είναι και αδύνατον από το ίντερνετ ή από το τηλέφωνο δεν έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίου. Παραδείγματο χάρη, οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι για τη διαδρομή Παρίσι-Μιλάνο δεν χρησιμοποιούν καθόλου πληροφορίες για όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες όπως το Βατερλό και συνιστούν τη χρησιμοποίηση αεροπλάνου. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ανεξάρτητο σύστημα πληροφόρησης στα e και στο ίντερνετ και το τηλέφωνο που να μιλάει για, όλους τους, για όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον επιβάτη και δεύτερον δεν πρέπει οι σταθμοί να την χάνουν εκμετάλλευσης μόνο από τις εταιρείε. Δεύτερον, σημείο της οδηγίας για το δικαίωμα των σιδηροδρομικών επιβατών πρέπει οι επιβάτες να έχουν το δικαίωμα επεξεργασίας πλήρως του ταξιδιού τους και να μην υπάρχει πληροφόρηση μόνο του σκληρού πυρήνα των πιο αποδοτικών γραμμών. Ξέρουμε βέβαια ότι ορισμένες εταιρείες αντιδρούν πολύ έντονα σε αυτό παρά το ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες για την εφαρμογή αυτού του σχέδιου. Τρίτη ιδέα δημόσιες υπηρεσίες και λειτουργική αποτελεσματικότητα. Φαίνεται ότι ορισμένες ιδρυμικές εταιρείες έχουν μια λογική αποτελεσματικότητας με βάση μόνο τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους που μπορεί να οδηγήσουν την κατάργηση ορισμένων υπηρεσιών που δεν είναι άμεσα αποδοτικές αντί να τις βελτιώσουν. Έτσι σε πολλές χώρες μειώθηκε η μεταφορά εμπορευμάτων αλλά και επιβατών ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός ο πληθυσμός. Η γαλλική εταιρεία, κρατική εταιρεία θα είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί όλες, όλη την επικράτεια αλλά τελευταία αποδείχθηκε ότι και η μείωση και η αύξηση της ε, μόλυνσης του περιβάλλοντος διευκολύνεται από τις ε, καταργήσεις ορισμένων γραμμών γιατί έτσι χρησιμοποιούνται περισσότερο τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Αυτή η λογική λοιπόν του άμεσου κέρδους δεν οδηγεί τελικά σε μείωση του κόστους από τις εταιρείε σε σύγκριση με την εποχή όπου υπήρχε μονοπόλιο. Και έτσι καταλήγουμε στην τέταρτη μας σύσταση το άνοιγμα στον ανταγωνισμό μεταξύ των συνδρομικών εταιριών για να υπάρξει μία προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και μείωση του κόστους. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι είναι δυνατόν και είναι προς το συμφέρον των επιβατών. Η πολλαπλότητα των εταιριών σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός των εποπτικών οργανισμών. Εμείς είμαστε υπέρ του ανταγωνισμού και όχι υπέρ του συνδυασμού και των μονοπωλίων. Και το δικαστήριο τελευταία μίλησε γι' αυτό στα πλαίσια της τέταρτης, σε συνδυασμό με την τέταρτη δέσμη. Η νομική ανεξαρτησία, η χρηματοδοτική ανεξαρτησία και η οργανωτική ανεξαρτησία, καθώς και στη λήψη αποφάσεων, είναι ουσιαστικά στοιχεία και προσθέτουμε ότι πρέπει να υπάρχουν και ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους. Η ευθύνη για τις υποδομές δεν είναι η ίδια η λογική του υπεύθυνου των υποδομών, δεν είναι η ίδια λογική με των σιδηροδρομικών εταιριών. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει ανεξαρτησία και των δύο. Αλλά αυτές οι δύο λογικές είναι και οι δύο απαραίτητες και συνδυάζονται. Η δημόσια υπηρεσία είναι κρατική και πρέπει να προβλέπει κρατική υποστήριξη. Όπως στη Γαλλία τα τρένα Intercity ή τα τρένα ΤΕΤ. E Πρέπει λοιπόν ορισμένες υπηρεσίες να ανατεθούν από τον κρατικό στον ιδιωτικό τομέα αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση τον δίκαιο ανταγωνισμό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζακό. Τώρα τα εθνικά ρυθμιστικά σώματα και υπηρεσίες, η κυρία Ήρις Χάνσελερ Ούγκε, αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Δικτύου της Γερμανίας. Ορίστε, κυρία Χάνσελερ Ούγκερ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πούμε ποιοι είμαστε. Εγώ εκπρόσωπο την ομοσπονδιακή, τον Ομοσπονδιακό ε, Οργανισμό Δικτύων ε, ε, μαζί με τις τηλεπικοινωνίες ε, και τη, τους σιδηροδρόμους από το 2006, τις υποδομές. Υπάρχει δίκτυο ανεξάρτητων σιδηροδρόμων που δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια. Υπάρχει κείμενο θέσεων για την τέταρτη δέσμη, αποφασίστηκε τέλος Απριλίου και οι ρυθμιστικοί φορείς της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας, της Γερμανίας συμφώνησαν 26 σε κείμενο θέσεων και καλύπτει και το θέμα της διακυβέρνησης. Είναι πολύ σημαντικό και να το διαβάσετε. Εγώ θα μιλήσω για την ε, εθνική αγορά επιβατών. Θα σας παρουσιάσω τη γερμανική εμπειρία Καταρχήν το άνοιγμα της ντόπια αγοράς μας βρίσκει σύμφωνους. Ανοίξαμε ήδη την αγορά στην Γερμανία και η εμπειρία μας είναι πολύ θετική. Έχουμε θετική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης της αγοράς και του ανταγωνισμού και της εξέλιξης των τιμών. Βλέπετε εδώ τα κομμάτια που έχουν ανταγωνισμό. Αυξήθηκε το μέγεθος της αγοράς και ε, μειώθηκαν οι τιμές. Επίσης ο αριθμός των υπηρεσιών ε, αυξήθηκε και το μερίδιο το σιδηροδρομικό αυξάνεται συνεχώς Οπότε η εμπειρία από τον ανταγωνισμό και το άνοιγμα των αγορών, της αγοράς στη Γερμανία είναι θετική. Επίσης ε, έχουμε κάποιες ανησυχίες σχετικά με το, τη, το, δοκιμή αυτή ε, ισορροπίας που μπορεί να ε, δημιουργήσει κάποια προβλήματα και μπορεί δηλαδή να είναι το αποτέλεσμα ένα κλείσιμο της αγοράς. Ε, τώρα, η υποχρεωτική ε, ανταγωνιστική διαδικασία διαγωνισμού ε, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και ποιότητα υπηρεσιών. Μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αυτή είναι η θέση του οργανισμού μας. Το μήνυμα είναι πολύ σαφές, αλλά τέλος βλέπουμε και ένα πρόβλημα γιατί η διαγωνιστική διαδικασία Γι' αυτήν δεν είμαστε εμείς ο αρμόδιος φορέας. Ε, τα κρατήδια είναι υπεύθυνα ε, και οι διαδικασίες ε, για τη διαδικασία ρυθμίζονται αλλού. Δεν υπάρχει να θεσπιστεί κάποιος άλλος φορέας που θα παρεμβαίνει και θα αναλάβει αρμοδιότητες εκεί. Τώρα για το unbundling, το διαχωρισμό εκμετάλλευσης ιδιοκτησίας, ε, αυτό συζητείται σε, όλου, σε όλους τους κλάδους δικτύων. Είναι παλιά συζήτηση αν θα διαχωρίσουμε δίκτυο και υπηρεσίες. Η θέση μας ε, είναι δεδομένη. Δεν λύνει τα πάντα ε, το unbundling. Εμείς ως οργανισμός θέλουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση προς το unbundling. Αν δούμε και την εμπειρία μας στις τηλεπικοινωνίες, λίγοι κανόνες unbundling ε, υπάρχουν, είναι ήπιοι, αλλά ο ανταγωνισμός λειτουργεί καλά, έχουμε μείωση τιμών, νέες διαδικασίες και επενδύσεις. Στην ενέργεια έχουμε κανόνες unbundling και σε αυτό το τομέα βλέπουμε εκπείρας ότι υπάρχουν και προβλήματα βέβαια, ε, έχει ε, πλεονεκτήματα το unbundling αλλά και προβλήματα ιδιαίτερα αν δείτε την αλλαγή στην ενεργειακή δέσμη στη Γερμανία υπάρχουν προβλήματα με το κόστος ε, συναλλαγών και τις συνέργειες αν έχουμε ολοκληρωμένους, ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ε, το πρόβλημα στην ε, οικονομική ισχύ ε, είναι κάτι που μας απασχολεί. Επίσης, όσο πιο ισχυρή η ρύθμιση, τόσο χαμηλότερο το επίπεδο, αναγκαίο επίπεδο unbundling. Επίσης, θα δείτε ότι υπάρχουν μονοπόλια και από το σκέλος της ζήτησης θα δείτε επιχειρήσεις σιδηροδρομικές που ε, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Οπότε είναι και οικονομικό το συμφέρον ε, παρά το unbundling. Και βλέπουμε ότι αυτό το μοντέλο εταιριών συμμετοχών μπορεί να συνεχιστεί και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός ε, αν είναι ισχυρός ο ρυθμιστικός φορέας και ανεξάρτητος. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει ε, οι ε, ρυθμίσεις ε, και το unbundling να μην είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, αλλά να αλληλοσυμπληρώνονται. Το νομικό πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές υποδομών θα δίνουν πρόσβαση στις υποδομές με διαφανή τρόπο, με αντικειμενική βάση, χωρίς διακρίσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε και ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα βάζει θεμέλια για ανεξάρτητους και ισχυρούς ρυθμιστικούς φορείς για να ε, πτυρούν αυτά τα δια, αυτές τις αρχές. Αυτό είναι σημαντικό και θετικό στο, στην τέταρτη δέσμη. Όμως ε, ε, υπάρχουν, πιστεύω, υπάρχει ο κίνδυνος το unbundling να προχωρήσει υπερβολικά ε, θα πρέπει να ισχύει στις μικρές υποδομές, δεν λύνονται με τον ίδιο τρόπο όλα τα προβλήματα. Επίσης ο έλεγχος της συμμόρφωσης του unbundling θα πρέπει να επικεντρώνεται στον ε, εθνικό, σε έναν ισχυρό ε, εθνικό ρυθμιστικό φορέα και να μην χωρίζεται μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Επίσης ε, η άρνηση της πρόσβασης φαίνεται να είναι αντιπαραγωγική ε, ως μέσον διασφάλισης συμμόρφωσης ε, με τους κανόνες του unbundling. Ο στόχος είναι το άνοιγμα, όχι το κλείσιμο της αγοράς. Και βέβαια θέλουμε να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις με διασυνοριακές δραστηριότητες. Οι κυρώσεις, αν οι κανόνες δεν πληρούνται ή πληρούνται εν μέρη, ε, θα πρέπει να εφαρμόζονται, αλλά πάντα πάνω στη βάση μιας, ε, ενός πλήρους ελέγχου ε, της, του τρόπου λειτουργίας τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Χένσελ Ούγκερ, πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις των βουλευτών, θέλω να καλωσορίσω What? Μια ομάδα από την, ε, τον ε, όμιλο τριανών που έφερε ο κύριος Ραμπράντμπον Καλώς ήλθατε και ελπίζω να είναι χρήσιμη αυτά που θα ακούσετε εδώ πέρα. Συζητούμε το συνδρομικό πακέτο. Φαντάζομαι ότι πολλοί από σας θα παίρνετε το τρένο και άλλα θα σας ενδιαφέρει. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Συνάδελφοι, έχω τους τρεις εισηγητές, Γκρός, Αλκαντράι, Κόλτσεκ, Πείτε ποιοι άλλοι θέλουν να μιλήσουν. Πέντε λεπτά θα έχουν το πολύ οι εισηγητές και τρία λεπτά το πολύ οι βουλευτές. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια μικρή διαπίστωση ε, έχοντας ακούσει τις απόψεις, διαπιστώνω ότι και εμείς δεν έχουμε νέα άποψη στο Κοινοβούλιο για την τέταρτη δέσμη μέτρων, για τις ιδεροδρομικές μεταφορές και εμείς και εσείς πρέπει να κάνουμε ακόμη πολλές συζητήσεις ε, για να πλουστεύσουμε τα πράγματα εδώ και τη διαδικασία της ακρόασης ε, τα σχόλια θα γίνουν ε, αργότερα. Ε, θα κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις μόνο. Καταρχήν στην κυρία Χένσλερ, ο ρυθμιστικός φορέας στη Γερμανία, δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να απαντήσετε, ελέγχει και την ροή ε, χρηματοδότησης ε, που θα πρέπει να καταβάλλονται και τα ε, κονδύλια που διατίθενται για τη βελτίωση του δικτύου γιατί συνολικά η χρηματική ροή ιδιαίτερα σε ολοκληρωμένες δομές είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα σχετικά σημαντικό θέμα γιατί μεταξύ άλλων προκύπτει ξανά και ξανά. Ε, επίσης, αν κατάλαβα καλά τον κύριο Ζακό, και αυτά που είπε για τους επιβάτες, δεν ξέρω, μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι το συμφέρον των εργαζομένων σε αυτό το τομέα διαφοροποιούνται από τα συμφέροντα των επιβατών, όπου οι τελευταίοι περιμένουν ότι θα είναι πιο αποτελεσματική μια διαχωρισμένη δομή, ενώ εσείς ως εκπρόσωποι των εργαζομένων πιστεύετε ότι οι ολοκληρωμένες δομές θα διατηρήσουν και θα προφυλάξουν τις θέσεις εργασίας καλύτερα. Ε, είναι σωστή η εντύπωσή μου αυτή, δηλαδή σαν να είναι ε, διαφορετικά εδώ τα συμφέροντα εργαζομένων και επιβατών. Ε, δεύτερη ερώτηση Ποια είναι η εξέλιξη της απασχόλησης του σιδηροδρόμους. Υποθέτομαι ότι τώρα η προστασία των εργαζομένων ήταν πιο έντονη, ενώ τώρα καμιά φορά αμφισβητείται. Επόμενη ερώτηση. Για τη, για τη διαχείριση της των υποδομών. Η ανεξαρτησία, αν κατάλαβα για καλά, είναι σημαντική για σας, όπως και η αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα των σιδηροδρόμων, που έτσι θα ενισχυθεί. Μπορεί να φανταστείτε και έναν ευρωπαϊκό διαχειριστή υποδομών που θα διαχειρίζεται μεγάλα δίκτυα, όπω ε, ε, ε, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα. θα ήθελα να μου πείτε πώς το βλέπετε, αν ε, αποτελεί θέμα για σας, πώς το προσεγγίζετε, γιατί αυτό βέβαια προϋποθέτει μία διαφορετική προσέγγιση ε, στη διαχείριση των υποδομών. Επόμενη ερώτηση προς τον ε, Λόρδο Μπέρκλεϊ. σάσα ε, σας ενδιαφέρει πολύ η, η επικερδής λειτουργία. Ο διαχωρισμός των, μεταξύ ε, ε, επιχειρήσεων και διαχειριστών είναι δαπανηρή, λέγεται. Πώς αντιδράτε σε αυτό, ότι ο διαχωρισμός δηλαδή μπορεί να αποτελέσει μια πολύ δαπανηρή πρόκληση. Κύριε Μωρέτη, εσείς βέβαια θέλετε μία ε, ήπια ολοκλήρωση των δομών των σιδηροδρόμων. Τι γνώμη έχετε σε σχέση με την προοπτική Ευρωπαίου ρυθμιστικού φορέα, γιατί αύριο αν θέλουμε να φτιάξουμε ευρωπαϊκό δίκτυο τότε η επιτήρηση δεν πρέπει να είναι ισχυρή μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά μεθαύριο θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προσεγγίσουμε το θέμα ε, μέσα από ευρωπαϊκή σκοπιά. Πώς βλέπετε το θέμα του ρυθμιστικού φορέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, μια ερώτηση στον κύριο Φόρστερ. Στην Αυστρία πόσο, πόσο χρόνο πήραν οι διαδικασίες με το ρυθμιστικό φορέα δηλαδή ε, είναι οικονομικά σωστό να λέμε ότι θα περιμένουμε μια απόφαση μετά από δύο χρόνια. Αν είναι βραδία η διαδικασία, μπορεί να ε, μην εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις. Επίσης, ε, έχει νόημα να γίνει προσφυγή είναι και ο, ο ρυθμιστικός φορέας είναι εκτός από ανεξάρτητος, αποτελεσματικός και ταχύς. Πέντε λεπτά, ο κ. Σαλκαντάουδη. Θα σας διαβάσω το κατάλογο των αγορητών για να υπάρχει και χρόνος για να απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας και μετά να μιλήσει και η Επιτροπή. Έχω Γκρός Καντράου, Κόλτσεκ, εισηγητές και κατόπιν. Mr. Zila, Mr. Ε, Kanchian, Mr. Benyon, Mrs. Durant, Mr. Eh, Savama, eh, Mr. Van Dalen and Mrs. Bilbao, Mr. Dibaka, Όσοι περισσότεροι μιλούν, αυτοί είναι μέχρι τώρα. Βλέπω σε ένα λόβα. Τελειώνω, κλείνω τον κατάλογο. Δύο λεπτά οι μη εισηγητές. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά και συγγνώμη για την πίεση. Κύριε Αλκαντράουι. Ευχαριστώ. Πρώτον, να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τη συνεισφορά τους. Οι διαφορές ε, των θέσεων αντικατοπτρίζουν σωστά τις δυσκολίες υλοποίησης της ε, διαδικασίες αυτή που νομίζω ότι είναι αναγκαίο τόσο και για τις εμπορευματικέ και για τις επιβατικέ μεταφορές. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να γνωρίσουμε τον στόχο μας, την νομοθετική μα δουλειά, που είναι να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό συνδρομικό σύστημα που θα είναι αποδοτικό, θα παρέχει ποιότητα και θα είναι θετικό όχι μόνο εκεί όπου υπάρχουν δυνατά κέρδη αλλά και σε γραμμές όπου οι μηχανισμοί της αγοράς δεν είναι πάντα υπανάκια. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών επιταγών που απαιτούν αποτελεσματικότητα και της προστασίας της δημόσιας υπηρεσίας και της προστασίας ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων στον κλάδο. Στον τομέα μου Συμβούλιο ε, Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας και Απελευθέρωση υπάρχει μια σύγχυση. Από τη μια μεριά μιλούν, ε, γίνεται λόγος για την ελεύθερη πρόσβαση όλων των φορέων και για την ε, διάσπαση των διαγωνισμών εκτός αν, όπως λέει η Επιτροπή, η οικονομική ισορροπία δεν, απολύ, δεν απειλείται. Τώρα, είναι παρκώς σαφές ε, αυτό το ε, σαφής αυτή η έννοια της ισορροπίας. Είναι δυνατόν να ανατεθεί μια σύμβαση και να γίνουν ε, ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της σύμβασης αυτής ή παράλληλα μπορούμε σε ένα-δύο χρόνια μετά να δεχθούμε ανταγωνιστές στην ίδια γραμμή. Σε μια τέτοια περίπτωση υπονομεύεται η βιωσιμότητα της πρώτης σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας. Και ρωτώ λοιπόν την κυρία, τον κύριο Φώστερ και τον κύριο Μωρέτη να μας διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε το κείμενό της ε, η Επιτροπή υπάρχει ο κίνδυνος ε, τα παλιά μονοπόλια να αντικατασταθούν από 3, 2, 3, 4 μεγάλα ολιγοπόλια. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι θετικό. Συμφωνείτε με την εκτίμησή μου. Ποια μέτρα κατά την πρέπει να ληφθούν τόσο στο μέλλον να υπάρχουν επαρκείς φορείς ποιοτικού χαρακτήρα στην Ευρώπη και όχι ένα ολιγοπόλιο. Τώρα, η άμεση ανάθεση έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη. Θα υπάρχει σχεδόν πάντα υποχρέωση δημόσιων διαγωνισμών. Ρωτώ, είναι η σωστή διαδικασία για κάποιες μικρές συμβάσεις πιο μεγάλες από αυτές που, παρέχει, που προτείνει το υφιστάμενο πακέτο δεν θα ήταν ίσως πιο σκόπιμο να έχουμε απευθείας ανάθεση. Τώρα για την ε, κοινωνική και εργασιακή διάσταση του θέματος λίγα μπορώ να πω. Οι προτάσεις της Επιτροπής, για τις προτάσεις της Επιτροπής θα καλούσα λοιπόν τους ε, προσκεκλισμένους μας, ιδίως δε τους νέου εισερχόμενους φορείς, τη Westbank, να μου πούν κατά πόσο συμφωνούν με τα συνδικάτα όταν, λένε πως ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες αμοιβών, η αγορά δημιουργούσε μία πίεση προς τα κάτω. Ερώτημα που θέτω και σε άλλους. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφευθεί αυτή η κίνηση της πίεσης προς τα κάτω, στους μισθούς ε, και στις συνθήκες εργασίας. Στον εκπρόσωπο της Westbank, οι δικοί σας εργαζόμενοι έχουν, δουλεύουν με τις ίδιες συνθήκες ε, ε, που έχουν και οι του κρατικού φορέα στην Αυστρία. Δομές για την κυρία Ένσλορ. Κύριε Ένσλορ, προτείνεται και προστατεύεται το γερμανικό μοντέλο, το καταλαβαίνω. Κατά την άποψή σα μια ένας θεμητός ανταγωνισμός μπορεί να γίνει με ενοποιημένες επιχείρησεις. Αλλά πέραν των εθνικών διαστάσεων υπάρχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Πώς δημιουργείται ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, δίκαιο, ε, δίκαιο ανταγωνισμό. Μια επιχείρηση όπως η δική στη Γερμανία δεν θα ήταν σε καλύτερη θέση αν θελήσει να ελέγξει άλλες επιχειρήσεις σε άλλα κράτη-μέλη. Για τον κύριο Μπέρκλεϊ μια ερώτηση. Οι, οι διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να ενισχυθούν εξού και ζητούμε διαχωρισμό μεταξύ διαχειριστή υποδομών και φορέα. Αλλά και για τη διεθνή διάσταση η φυστάμενη νομοθεσία προβλέπει διαδρόμους διεθνείς ε, διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών. Λειτουργούν αυτά ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει στο νέο πακέτο κάποιας ε, συμπλήρωση για να υπάρχει, είναι, για να υπάρχει καλύτερος συντονισμός. Κύριε Κόλιτσεκ. Ναι, οι και μετά όλοι γιατί αλλιώς Μιχάλη δεν θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Κόλιτσεκ λοιπόν. Ευχαριστώ. Τους άκουσα όλους πολύ προσεκτικά και κανείς δεν είπε ότι η αποσύνδεση βελτίωσε τη λειτουργικότητα, ιδίως για τους επιβάτες. όταν αντί για ε, μία εταιρεία υπάρχουν 8, μειώνεται η αποδοτικότητα, η λειτουργικότητα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αρχίσα, άρχισε η αποσύνδεση με η τελεία καταστροφή και τώρα αρχίζει να βελτιώνεται κάπως η κατάσταση. Κατά τα άλλα, όπως μας έδειξε και το παράδειγμα της Bundesmann, ορισμένα δρομολόγια όπως Βιέννη Λίντς μπορεί να είναι αποδοτικά με πολλαπλές εταιρείε, αλλά τα υπόλοιπα δεν είναι οικονομικά ενδιαφέροντα. Εκτός αυτού, συμφωνίες Οποιασδήποτε συμφωνίες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλα τα δρομολόγια, όχι μόνο τα κύρια αλλά και τα λιγότερο αποδοτικά. Ποιος θα πληρώσει για τα δεύτερα αυτά. Θα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος και λιγότερη ασφάλεια. Τέλος, τα δρομολόγια δεν είναι άπειρα. Σε πολλές χώρες υπάρχουν δυνατότητες για σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, σε άλλες όχι. Στη δική μου περιφέρεια προβλέπεται κατάργηση πολλών δρομολογίων. Και θα ήθελα να πω ότι αν εφαρμοστεί ο δικαίος έχει, τότε, τότε λέγω, ιδιαίτερα τα εθνικά δρομολόγια θα επηρεαστούν και η αποζημίωση που προβλέπεται δεν θα υπάρχει πια. Ούτε θα υπάρξει άλλη αντιστάθμιση και δεν θα ήταν καλό να μείνουν τα πράγματα έτσι. Κάτι ακόμα, το σημείο 63 της αναθεώρησης του, της πρώτης δέσμης λέει ότι η Κομισιόν θα κάνει πρώτα μια ανάλυση και μετά θα ληφθούν μέτρα. Πώς γίνεται όμως η Κομισιόν να μην έχει ακόμη σεβαστεί αυτή την υποχρέωσή της από την πρώτη σιδηροδρομική δέσμη. Και τώρα επεξεργάζεται κάτι τελείως διαφορετικό που παραβιάζει όλους τους ισχύοντες κανόνες. Έπειτα το 63 λέει επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές. Ακόμη μια φορά λοιπόν η Κομισιόν ερωτώ γιατί δεν σέβεται την υποχρέωση που είχε αναλάβει. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα η ανάλυση που προβλέφθηκε από την προηγούμενη δέσμη. Το recast από την πρώτη δέσμη δεν εφαρμόστηκε η ανάλυση του τουλάχιστον των αποτελεσμάτων και πολλές χώρες είχαν σοβαρούς λόγους για να μην την εφαρμόσουν. Πώς μπορούμε να δεχτούμε ότι θα υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες στις διάφορες χώρες, αλλά ταυτόχρονα θεωρούμε ότι είναι ένα ενιαίο σύστημα καλό. Τότε γιατί δεν εφαρμόζεται παντού. Υπάρχουν λοιπόν χώρες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέλη. Μιχαήλ, δύο λεπτά για σένα ως εισηγητής θα έχει το απόγευμα πέντε λεπτά και θα έχουν οι άλλοι δύο λεπτά. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όλους τους ομιλητές. Ναι, αλλά παρόλα αυτά συνήθως οι συντονιστές έχουν περισσότερο χρόνο από τους άλλους. Είναι άδικο. Να μιλήσουν περισσότερο οι συντονιστές, αλλά τότε θα πρέπει τα υπόλοιπα μέλη, ο κυρίος και η κυρία Ντουράντ, ε, θα έχουν λιγότερο χρόνο. Ευχαρίστως να πάρουν τρία λεπτά οι συντονιστές, αλλά οι άλλοι θα έχουν λιγότερο χρόνο. Και οι φιλελεύθεροι θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο δικός τους ο συντονιστής τότε. Τρία λεπτά λοιπόν θα πάρεις εσύ και θα ε, τρία λεπτά οι φιλελεύθεροι και ο κύριος Σέλερ τρία λεπτά. Βλέπετε, αρχίζουμε τα, τις διαφωνίες. Τρία λεπτά λοιπόν ο Μίχαελ. Λοιπόν, για το cherry picking, τις επιλογές κάποιων, οι Σκιώδης, δύο λεπτά. Η απόφαση ελήφθη. Μίχελ. Τώρα, για το cherry picking. Το cherry picking δεν είναι πρόβλημα αν, ας πούμε, έχουμε τέσσερις σειρμούς σε μία ώρα κάθε 20 λεπτά και μετά δύο ώρες χωρίς άλλο σύρμο. Ε, θα υπάρξει άλλη ρύθμιση και συντονισμός. Γίνεται αυτό στη Γαλλία, αλλά οι περιφέρειες δεν το λαμβάνουν υπόψη. Ο πελάτης πρέπει να είναι στην πρώτη θέση. Τώρα, η κυρία Τρίερ. Αν υπάρχουν ελάχιστοι μισθοί, τότε αυτό που λέτε δεν ισχύει. Εμείς τους ελάχιστους μισθούς τους ε, θέλουμε. Ε, και αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση. Και βεβαίως δεν θέλουμε κοινωνικό dumping. Ε, τώρα οι τιμές ε, αυξάνονται πολύ για τις γραμμές και πώς, αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε κυρία Χέντζλερ την αύξηση τιμών. Κύριε Μωρέτια, από το Μόναχο στη Βενετία σε ορισμένους σταθμούς δεν σταματούν. Μετά το Μιλάνο μόνο σε ορισμένους. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Πώς, τι κάνετε γι' αυτό. Τώρα τα εισιτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπαμε ότι είναι ε, ε, ρυθμισμένο το θέμα, δεν εφαρμόζεται όμως. Πώς θα δημιουργήσουμε ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο αφού δεν έχει ρυθμιστεί αυτό. Επίσης, κυρία Χάντσιλερ, τι κάνετε σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δεν θέλουμε τρία ολιγοπόλια, εγώ είμαι κατά των μονοπωλίων ιδιωτικών ή κρατικών, αλλά αν οι ρυθμίσεις μας σημαίνουν ότι θα έχουμε μονοπόλια που υπαγορεύουν κανόνες στην αγορά, τότε χάνεται και από εκεί ο ανταγωνισμός. Επίσης το Ζάξεν Άνχαλ, το Deutsche Bahn είπε ότι αν υπάρξουν αυξήσεις ε, αυτές δεν θα τις αναλάβουμε εμείς, θα κινηθούμε μόνοι μας και έχουν ένα πλεονέκτημα. Αυτό είναι μεγάλη διάκριση. Ποια είναι η θέση σας ε, εδώ. Επίσης λέτε ότι οι αρχές εθνικές και ευρωπαϊκές πρέπει να συνεργάζονται. Σωστό και συμφωνώ και εγώ, αλλά ποιος έχει τον τελευταίο λόγο, η εθνική αρχή ή η ευρωπαϊκή το, στο 95% των περιπτώσεων δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Αλλά αν υπάρξει σύγκρουση, πιστεύω ότι η, Ευρωπαϊκή Αρχή πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο. Τέλος, ε, ότι δεν ε, δίνει τίποτε ο ανταγωνισμό. Ήμουν εισηγητή στην πρώτη δεσμή μέτρων και είδαμε ότι αυτοί που άνοιξαν την αγορά στις εμπορευματικέ μεταφορές ε, από χαμηλότερο επίπεδο, η Μεγάλη Βρετανία συν 60%, συν 30% η Πολωνία και ε, στη, Γαλλία, στη Γαλλία έχασαν 25%. Ερωτώ λοιπόν και εσάς, αυτές είναι απώλειες θέσεων εργασίας ε, μετά από αυτά που έγιναν και αν είστε κατά του ανταγωνισμού πρέπει αυτό να το λάβετε υπόψη σας. Και στις ε, ε, επιβατικές μεταφορές ε, στον Düsseldorf Μέτμαν θέλαν να σταματήσουν τη γραμμή γιατί ήταν μόνο 500 επιβάτες κάθε μέρα. Το ανέλαβαν ε, ανταγωνιστές ιδιώτες και τώρα ανέβηκε ο αριθμός των επιβατών στις 23.000. Αυξήθηκαν λοιπόν τώρα αυξήθηκε και ο αριθμός των θέσεων εργασίας. λοιπόν, πώς βλέπετε αυτό το θέμα που λέτε ότι που δεν πρέπει να έχουμε ανταγωνισμό. Ο κύριο Ζήλερ, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις όλους ε, τους ε, προσκεκλημένους μας. Μία ερώτηση προς όλους. Έχουμε όλους παρόντες. Ποια είναι η αποψή σας. Το πακέτο πρέπει να μείνει πακέτο ή να χωριστεί. Γιατί είδα και κάποιες αντιφάσεις που ε, αντιρρήσεις που ακούστηκαν. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό. Έπειτα, την κυρία Τρίρ, αναγνωρίζω ότι τα συνδικάτα έχουν πολύ σημαντικό πολιτικό ρόλο. Είπατε ωστόσο ότι σας πλήττει η νέα νομοθεσία. μέσω ή μακροπρόθεσμα αυτό είναι λάθος. Λέτε ότι είσαστε κατά της, ε, του κατακαιρματισμού των επιχειρήσεων στον τομέα. Ταυτόχρονα θέλετε να κρατήσετε ωστόσο τον κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας. Δεν ξέρω πόσα μέλη των σιδεδομικοί είναι μέλη των οργανώσεών σας, αλλά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των μελών σας και μισθολογικά και εργασιακά. Στην το βλέπουμε και σε άλλους κλάδους του, σε αεροπορικές μεταφορές. Οι πιλότοι, ας πούμε, δουλεύουν πανευρωπαϊκά μόνοι τους. Και η ερώτηση που θέτω είναι, μακροπρόθεσμα η σιδηροδρομικοί θα πρέπει να, απαντήσουν στο εξή δίλημα. Πιο ανταγωνιστική σιδηρόδρομη με καλύτερους μισθούς εν τέλει για τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους ή έναν κατακαιρματισμένο ψηδομικό κλάδο που χάνει στις μεταφορές και κανένα μέλλον για τους εργαζόμενούς του. Κύριος Ντιμπάκε, για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσεις των προσκεκλημένων μας. Εγώ διαπιστώνω ότι όλες ε, παρεμβάσεις με την εξαίρεση της εκπροσώπου των συνδικάτων είδαν το πακέτο με θετικό τρόπο. Αν επιτρέψει το άνοιγμα των αγορών και βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών για τους επιβάτες είναι κάτι το θετικό. Οι φιλελεύθεροι πάντα θεωρούσαν ότι το άνοιγμα της αγοράς ήταν κρίσιμο. Όσο περισσότεροι φορείς υπάρχουν στην αγορά, τόσο καλύτερες θα είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους επιβάτες. Γι' αυτό και κατά την άποψή μου, ο χωρισμός είναι αναγκαίος, απαραίτητος, ούτως ώστε οι διάφοροι φορείς να μπορούν να μπουν στην αγορά σε ένα level playing field ισότιμο επίπεδο για όλους, με καλύτερο συντονισμό. Και η πλατφόρμα θα επιτρέψει να έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι με ισότιμο τρόπο στην αγορά. Η ερώτησή μου προς τη Γερμανία, εκπρόσωπο του, της γερμανικής ρυθμιστική αρχή, Τι θα κάνει αν δεν γίνει πλήρω κάθε, ο κάθετος διαχωρισμό, διότι μπορεί να έχει χρηματοοικονομικέ χρηματοοικονομικές και ροέ προσωπικού που θα δώσουν στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Πώ θα γίνεται λοιπόν στην πράξη ο έλεγχο. Εγώ έχω μια λογιστική εμπειρία και μπορώ να σα πω ότι λογιστικά μπορεί να γίνουμε πολύ δημιουργικοί. Πώ θα το ελέγχετε λοιπόν αυτό. Μια τρίτη ερώτηση προς, τους ε, προς τον εκπρόσωπο των επιβατών. Είδατε την πρόταση επιτροπής με θετικό τρόπο. Τι θέλετε ωστόσο συμπληρωματικά στην πρόταση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε βελτίωση της ποιότητας που παρέχεται στον επιβάτη. Και τρίτον, στους ε, φορείς και διαχειριστές των υποδομών. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει πλήρης χωρισμός υποδομών και ε, δικτύου. Α το υποθέσουμε. Κάπου σε κάποιες χώρες τη Ευρώπη αυτό συμβαίνει. Μήπως διαπιστώσουμε τότε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες τους ώστε το κόστος των ε, συναλλαγών που σχετίζονται με, την, ε, ε, με το διαχωρισμό λύνονται μέσω μιας προσέγγισης πλατφορμικής που θα οδηγήσει σε μια στενή συνεργασία ίσως και ενσωμάτωση και θα επιτρέψει η δημιουργία οικονομιών κλίμακας όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό πώς το βλέπετε. Euh, Κυρία Ντουράν, ευχαριστώ. Να πω στον εκπρόσωπο του ΣΕΡ ότι Συμφωνώ μαζί σας ότι το κείμενο της Επιτροπής προσανατολίζεται πολύ σε, συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και να πω και στον κύριο Μπρέκ, δείτε την ανάλυση που είναι λεπτομεριακή και συγκριτική ανάλυση της απελευθέρωσης του κλάδου στην Βρετανία και θα δείτε ότι παρότι υπάρχει 60% αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών υπάρχει και μία ε, εικόνα αποκάλυψης ταυτόχρονα και αυτό το γράφει κάποιο που είναι υπέρ τη απελευθέρωση Δεύτερον, Στου εκπροσώπους των επιβατών θα έχετε τι ενοποιημένες υπηρεσίε που περιμένετε ή είναι εφικτό κάτι τέτοιο αν σπάσουμε τελείως τις επιχειρήσεις. Και εγώ δεν μιλώ μόνο για τον έλεγχο του ανταγωνισμού αλλά και για την ποιότητα τη λειτουργία και τη δουλειά. Αν σπάσετε τι επιχείρησει δεν θα έχετε ενοποιημένη υπηρεσία. Τρίτον, πάμε βεβιασμένα, πολύ γρήγορα, με ένα κακό ακτιμημένο κείμενο. Δεν ξεκινήσαμε το 63 του Recast που ζητάει αξιολόγηση πλήρη με βάση την υφιστάμενη κατάσταση. Δεν έχουμε χρόνο καν να εφαρμόσουμε το Recast και έχετε ένα τεράστιο συμπληρωματικό Big Bang το οποίο δεν ξέρω αν θα, θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Διαπιστώνω λοιπόν μεταξύ σας πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις αλλά και όπως και σε εμά για το κατά πόσον είναι σοβαρό το νέο κείμενο και αν η αξιολόγηση έχει γίνει ε, με το σωστό τρόπο αλλά και για τους τρόπους για την υλοποίηση της ε, αλλαγής αυτής που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες δυσκολίες για τους επιχειρηματίες. Ευχαριστούμε. Κάντια. Κύριε Σκαντσιάν, ευχαριστώ. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία φορά αυτή που θα μιλήσουμε για πακέτα σιδηροδρομικών μεταφορών. Ελπίζω ότι η πρόταση που μας υποβάλλεται θα ενισχυθεί με τη δουλειά μας, γιατί και εγώ είμαι πεπισμένος ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε κάτι τέτοιο. Τα βασικά στοιχεία είναι οι κανόνες που πρέπει να, είναι, να μείνουν σταθεροί και οι πόροι που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Πώς θα βρούμε τους πόρους, πώς θα γίνουμε πιο ελκυστικοί. Μην ξεχνάτε ότι το να μιλάμε για νομοθεσία που εφαρμόζεται το 2019 και 2023 όπως κάναμε στο, στο αναδιατυπωμένο κείμενο δεν νομίζω ότι αποτελεί καλή πολιτική από τις παρεμβάσεις που έγιναν, εγώ θα έκανα μία βασική, ε, θα έλεγα ένα βασικό θέμα. Καταρχάς, για τον κύριο Μωρέτη, από την εμπειρία του. Ποιες προτάσεις θα μπορούσαν να καταστήσουν πιο ορατό για μας το συνδεδομικό πακέτο και να είναι και πιο ελκυστικό για τις επενδύσεις. Για τις ε, βασικές προϋποθέσεις. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή. Είναι αλήθεια ότι οι βασικές συνθήκες δεν είναι σωστές, πλήρεις και δεν έχουν τη, διάσταση, τη σωστή διάσταση, γιατί αυτό θα, θα έκανε την πρόταση πιο προβληματική. Τρίτη ερώτηση προς την κυρία Ένσλερ. Ασχολείται με τους εργαζόμενους. Μπορείτε να με πείσετε κάπως περισσότερο ότι ένας ισχυρός, μια ισχυρή ευρωπαϊκή ή εθνική ρυθμιστική αρχή θα εμποδίσει το ή θα δώσει εναλλακτική λύση στο unbundling. Εγώ χρειάζομαι μεγαλύτερη, να πιστώ περισσότερο. Γιατί για την απελευθέρωση είμαι απόλυτα βέβαιο και ότι πρέπει να υπάρξει και με αμοιβαιότητα. Για το unbundling μου δημιουργήσετε κάποιες ε, αμφιβολίε. Πείστε με ότι υποκαθίσταται από σωστή ρυθμιστική αρχή. Τελευταία παρατήρηση, πρόεδρε. Στην Ιταλία Είχαμε το NTU που ήταν ο μόνος Ευρωπαίος που έκανε ε, ανταγωνισμό. Ε, μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η εμπειρία αυτή δεν είναι ανήθικη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ανοιχτά. Δεν ε, μου αρέσει τόσο πολύ να μιλώ για τα θέματα αυτά, ε, στη και γραμμές κλπ. Έχω συμμετάσχει σε τέτοιες ακροάσεις και βλέπω πάλι τα ίδια πράγματα. Γίνονται καταγγελίες, αναφέρονται απειλές, αλλά δεν μιλάμε για ε, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών. Κανείς δεν λέει ότι θα ήταν καλό και λογικό να σκεφτούμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ε, πολύ λίγο συζητούμε για όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Μπέρκλεϊ, ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε, αλλά μεταξύ άλλων είπατε ότι θα υπήρχε αύξηση 60% υπήρξε 60% αύξηση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, πώς τα καταφέρατε. Βέβαια, εντάξει, μπορώ να διαβάσω αυτά που ε, γράψατε και ετοιμάσατε, αλλά πείτε μας κιόλας εδώ στην ακρόαση. Τώρα για τον οργανισμό δικτύων εσείς πρέπει να φροντίζετε για τη σωστή κατανομή των γραμμών κλπ. Πώς θα το ε, κάνετε αυτό και πώς θα το διασφαλίσετε. Ε, αν ας πούμε έρθουν οι Ολλανδοί στη Γερμανία και πούν ότι θα κινηθούν και Ολλανδικοί σύρμοι, πώς θα υπάρχει ε, δίκαιη πρόσβαση στο δίκτυό σας που δεν θα ευνοεί την Deutsche Bahn. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλεν. Η ε, κυρία Σενάλοβα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Μας είπατε πολλά πράγματα και δεν προλάβατε να μιλήσετε για την ασφάλεια. Θα ήθελα να ακούσω αυτό το κομμάτι της ε, ομιλίας σας. Θα μας απασχολήσει το θέμα το απόγευμα βέβαια, αλλά πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι μπορούν ε, κάλλιστα να μιλήσουν για την ασφάλεια. Τέλος, κάτι που εν μέρη επίσης αναφέρθηκε εδώ, η μετά ε, τη θέση σε ισχύ της ε, οδηγίας ε, θα διατηρηθεί το μοντέλο των εταιριών συμμετοχών. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις και μία ερώτηση στον κύριο Μπέρκλη. Όπως ακούσαμε από τη συζήτηση, ε, το Κοινοβούλιο δεν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο για όλα αυτά. Και η συζήτηση αποκαλύπτει επίσης πόσο δύσκολο είναι για το κοινοβούλιο μας να εξετάσει την γνήσια απελευθέρωση των αγορών. Άκουσα κάποια περίεργα πράγματα να λέγονται εδώ. Μιλήσαμε πολύ για τους επιβάτες. Προσθέτω κι εγώ ότι θεωρώ ότι ο επιβάτης είναι ο βασιλιάς και αν θέλουμε γνήσια απελευθέρωση της αγοράς τότε οι επιβάτες θα είναι ικανοποιημένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει κάτι που ξεπερνά του χειρότερους εφιάλτες σας. Προτείνει απλώς ότι το άνοιγμα των αγορών μεταφορών επιβατών θα γίνει μόνο σε αγορές που έχουν πάνω από ένα ελάχιστο μέγεθος. Μην φοβόμαστε τόσο πολύ λοιπόν. Επίσης ε, για την κυρία Τρίερ παρουσιάσατε την απελευθέρωση ως ε, φρίκη. Ε, ποιοι είναι οι καλύτεροι εργοδότες είναι αυτοί που έχουν επιτυχημένες εταιρείες και έχουν καλή θέση στην αγορά. Αυτοί φροντίζουν περισσότερο τους εργαζομένους. Και περνάω στην ερώτηση του κύριο Μπέρκλεϊ. Είπατε, και συμφωνώ ως επιτοπλίστων μαζί σας, είπατε τέλος πάντων ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τεχνικά ή νομικά εμπόδια που θα επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη και ότι όλα θα πρέπει και θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός γραμμών, πλήρης διαλειτουργικότητα. Μετά όμως είπατε, εκτός και αν σε κράτος μέλος υπάρχει απόλυτη ανάγκη για ειδική ρύθμιση. Καλό θα ήταν αν έχουμε χρόνο να το εξετάσουμε αυτό τι εννοείται, ποιες είναι αυτές οι απόλυτες ανάγκες που μπορούν να προκύψουν σε κάποια κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάνιον. Να επανορθώσω κάποια αρνητικά σχόλια για το βρετανικό σύστημα. Μετά την ιδιωτικοποίηση, στο, στο Στάφορσιρ, ο τοπικός σταθμός έχει τέσσερα τρένα για το Λονδίνο κάθε μέρα και κάθε δύο ώρες ένα για τον Birmingham. 18 χρόνια αργότερα έχει κάθε μισή ώρα στο Birmingham και κάθε χρόνο στο Λονδίνο και αυτό εξηγεί πολλά. Ε, είναι χαρακτηριστικό για όλη τη χώρα. Εξηγεί και την, ε, ε, το συνοστισμό που βλέπουμε. Οι ερωτήσεις μου αφορούν την εκπρόσωπο των συνδικάτων, και δεν βλέπω τα ονόματα και δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου, γι' αυτό συγγνώμη που δεν λέω το όνομά σας. Δεν κατάλαβα, είστε κατά της δημιουργίας ενιαίου χώρου σιδηροδρόμων ή όχι. Φάνηκε ότι είστε κατά του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου σιδηροδρόμων. Αλλά πώς μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικούς σιδηροδρόμους ε, αν έχουμε αυτή τη θέση. Επίσης από το, τη ρυθμιστή, την εκπρόσωπο ε, γερμανικής, της Γερμανικής Ρυθμιστικής Αρχής θέλετε κάποιο υβριδικό σύστημα μεταξύ διαχωρισμού και ενοποίησης ολοκλήρωσης και πώς θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Έχετε συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή μια επιχείρηση θέλει να είναι σιδηροδρομική και που λέει αυτό το κομμάτι είναι ενοποιημένο» και τότε θα πρέπει να αναλάβουμε, να το κάνουμε προσφορά στο διαγωνισμό και για την υποδομή. Α, αυτό είναι ένα αξιόπιστο μοντέλο. Και επίσης ε, και ο Τόνι Μπέρκλεϊ τι πιστεύει για το συγκεκριμένο ερώτημα. Τόνι, επίσης, ποια είναι τα βασικά εμπόδια για την δημιουργία ε, μια αγοράς μεγαλύτερης, διευρωπαϊκή για τους Ναύλου, Φταίει το, τα, φταίνουν τα προβλήματα ανοίγματο αγορά ή είναι τα προβλήματα που θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα. Και ποιο ήταν ο αντίκτυπο σε σχέση με συνθήκε εργασία και αριθμό απασχολουμένων στι χώρε που ε, προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση. Ζουρίμι, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ όλους τους ομιλήσαντες ομιλητές, όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα λειτουργικό διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά είναι δύσκολη η εφαρμογή του φαίνεται. Από αυτά που είπε ο κύριος Μωρέτη δεν τα κατάλαβα όλα, γιατί μας είπε ότι οι μελέτες αξιολόγηση της Κομισιόν δεν είναι αντικειμενικές. Είναι δυνατόν να γίνει μια υγιή, σωστή και σαφή συζήτηση με βάση μελέτες που να είναι προσανατολισμένες πολιτικά. Εγώ νομίζω ότι ως βουλευτές χρειαζόμαστε αντικειμενικότητα. Η Κομισιόν λοιπόν μπορεί να αναλάβει νέες μελέτες όπως τη ΣΕΡ που αναφέρατε. Γιατί ο κύριος Μωρέτη μας λέει ότι οι υπάρχουσες μελέτες δεν είναι σωστές. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μελέτες που δεν θα είναι σωστές και που χρησιμοποιούνται από συμφέροντα. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που θέτω είναι, με βάση αυτά που είπε ο κύριος Μωρέτη, μπορούν να υπάρξουν άλλες μελέτες εκτός από τις Κομισιόν. Κύριε Μπάρκλη, μας λέτε να σεβαστούμε τους κοινούς κανόνες για να υπάρξει ανοιχτή αγορά. Προφανώς έχετε δίκιο. Ερωτώ όμως, ο σεβασμός των κοινών κανόνων σημαίνει ενιαίο και επιβαλόμενο και υποχρεωτικό πρότυπο διακυβέρνησης. Περίεργο για ένα φιλελεύθερο να ζητάει την επιβολή ενός ενιαίου μοντέλου, ενώ σήμερα ζητιέται η συμμετοχή. Τέλος, με εκπλήσει ότι μόνο η εκπρόσωπος των συνδικάτων αναφέρθηκε στα κοινωνικά. Είναι πολύ ενισχυτικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν μήπως και οι άλλοι να μας διαβεβαιώσουν ότι και εκείνοι ενδιαφέρονται για το κοινωνικό συμφέρον των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους. Θα ήθελα να μου απαντήσει ο καθένας. Ευχαριστώ. Ξεκινώ λέγοντας ότι συμφωνώ απόλυτα με την δήλωση της Μόνικα Χέμινγκ που αν ξανακούσω πακέτο θα πάω σπίτι μου. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι ξέρουμε τα προβλήματα που έχει το άνοιγμα της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουμε γιατί δεν εφαρμόστηκε πλήρως το τρίτο πακέτο και όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Ως νομοθέτες τη στιγμή που υποβάλλουμε τις προτάσεις και πρέπει να τις προσπίσουμε στα μεγάλα, στους μεγάλους ομίλους ε, που, και τις δυσκολίε που έχουν τα κράτη να εφαρμόσουν το πακέτο. Νομίζω λοιπόν ότι ξεκινώ από το ότι όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ρωτώ λοιπόν τους προσκεκλημένους μας. Εφόσον θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό συνδρομικό δίκτυο, τι ρόλο πιστεύετε ότι πρέπει να παίζει ένας Ευρωπαίος ρυθμιστής, μια Ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Ποιος θα ήταν ο ρόλος του και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Αυτό είναι κομβικό ερώτημα αν θέλουμε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ε, διακυβέρνησης ή όχι. Με σαφή και λιτό τρόπο θα ήθελα να έχω την άποψή σας. Επίσης, να πω στην κυρία Τρίλ ότι πιστεύω πως το άνοιγμα της αγοράς, τα παραδείγματα τουλάχιστον που δείχνει, είναι ότι αν βελτιώσουμε την ποιότητα και τις υπηρεσίες, μπορούμε να βελτιώσουμε και την κατάρτιση των επαγγελματιών. Επίσης, το άνοιγμα της αγοράς θα είχε και δυνατότητες μεγαλύτερης καινοτομίας και βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού στον κλάδο. Με αυτή τη σύντομη παρέμβαση νομίζω σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάο. Θα επανέλθουμε τώρα στους ομιλητές με τη σειρά με την οποία μίλησαν από τον κύριο Φόρς μέχρι την κυρία Χένσλε Ρούγκε. Και λόγω του χρόνου θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε μόνο στα ερωτήματα που σας τέθηκαν και όχι να μην αναφερθείτε σε γενικότητες. Τρία λεπτά ο καθένας. Και αυτό είναι το ανώτατο, δεν είναι ανάγκη να μιλήσετε τρία λεπτά. Ο κύριος Φώστερ πρώτος. για τις ρυθμιστικές διαδικασίες και τη διάρκεια μεταξύ δύο μηνών και ενός έτους. Τώρα, αν οι προσφυγές έχουν νόημα. Όχι, ελάχιστο. Έτσι κι αλλιώς είναι δαπανηρή διαδικασία. Στην αρχή το κάναμε και άρχισαν μακρές διαδικασίες. Στην Αυστρία θεωρούμε ότι η ρυθμιστική αρχή είναι ανεξάρτητη και έχουμε και πολύ καλή εμπειρία από την ρυθμιστική αρχή που, λαμβάνει, που βοηθάει να λαμβάνονται ανεξάρτητες αποφάσεις που αλλιώ δεν θα ήταν δυνατόν να ληφθούν. Ο κύριος Κατράου ρωτάει σε ποιο βαθμό αντικαθιστούν τα ολιγοπόλια, τα μονοπόλια. Αν δούμε την πρόταση της Κομισιόν σε σχέση με τους ε, διαγωνισμούς, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί που μπορούν να ε, συμμετέχουν και το σύστημα γίνεται πλουραλιστικό. Δεν θα πάθει ζημιά το σύστημα. Αφενός έχουμε επιχειρήσεις σε ε, διαδρομές που ε, λειτουργούν χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς αύξηση για τους ε, ε, πολίτες και έχουμε και τους διαγωνισμούς που αντικαθιστούν τις απευθείας αναθέσεις και αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός ρίχνει τις τιμές για τις επιχειρήσεις και τους αναθέτοντες και υπάρχει θετική εξέλιξη με την τέταρτη δέσμη μέτρων δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν ε, ρίχνουν στη μέση οι διαγωνισμοί, όπως στη Βαβαρία, για παράδειγμα, όπου έδιναν λιγότερα χρήματα και είχαν μεγαλύτερη ποιότητα και αύξηση των μεταφορών, ε, μπορούμε να δούμε ότι αυτό το σύστημα θα βελτιώσει και τις τοπικές μεταφορές, θα τις πυκνώσει. Σε τρία λεπτά δεν θα προλάβω να τα απαντήσω όλα, αλλά ε, να πω κάτι για τον κύριο Κόλιτσεκ. Δεν συμφωνώ ε, με αυτό που είπε. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή να μην προωθεί πια απευθεία αναθέσεις, αλλά να τις αντικαταστήσει με διαγωνισμούς για να τονώσει τον ανταγωνισμό. Εμείς ε, θέλουμε να ε, τους διοργανώνουμε όμως με βέλτιστο τρόπο. Επίσης, ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ε, συνεργάτες μας, τους εργαζομένους. Εμείς δουλεύουμε με βάση συλλογικές συμβάσεις ε, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, του ιδιωτικού σιδηροδρόμους. Προβλέπεται και κατάρτιση. Το Υπουργείο παρακολουθεί τις δραστηριότητές μας και είναι απόλυτα ικανοποιημένο Δηλαδή ε, ο ανταγωνισμός και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, δεν ε, υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ούτε την ασφάλεια. Και στο τέλος έχουμε με αυτόν τον τρόπο ικανοποιημένους πελάτες. Ευχαριστώ. Μπορεί να απαντηθούν οι ερωτήσεις και με email αν κρυθεί σκόπιμο εδώ από το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μωρέτη, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για την πρώτη ερώτηση. Οι βάσεις για να αποφύγουμε μακρές ε, απαντήσεις ε, φροντίσαμε στα γραμματοκιβώτια όλων των ε, βουλευτών να υπάρχει σύνοψη της μελέτης που σας ανέφερα. Και όλη η ακαδημαϊκή μελέτη με 53 ερωτήματα για το impact assessment. Οπότε θα ελέγξουμε τα προβλήματα εν γέννη με πολύ εφαρμοσμένο τρόπο όλα τα θέματα. Δεύτερο θέμα, το cherry picking. Η επιλογή δηλαδή των καλύτερων ε, διαδρομών. Αυτό πρέπει να λυθεί το θέμα, είναι θέμα που πρέπει να λύσει η πολιτική. Εγώ σας έδωσα παραδείγματα στην Ιταλία με την NTU. Είναι προφανές ότι κάθε επιχείρηση και η incumbent σε ένα σενάριο που απελευθερώνει τις ε, μεταφορές βάσει του cherry picking πάει εκεί που υπάρχουν λεφτά και τα αφαιρεί από εκεί που χάνει λεπτά. Με το NTV στο στα υψηλής ε, ταχύτητα στρένα της Ιταλίας μειώνουν ε, κατά 100 εκατομμύρια τα profit. Τι τα έκανα αυτά τα χρήματα πριν για να τα χρησιμοποιούσα για να καλύπτω τις απώλειες, τις ζημίες στη γραμμή της Ευρετικής και του Τυρινικού. Και τι έκανα τώρα, έκοψα τα τρένα. Άρα έχουμε 60% προσφορά μεγαλύτερη από την ζήτηση μεταξύ ημών και του ανταγωνιστού στην κεντρική γραμμή, ενώ στις άλλες δεν υπάρχουν τρένα. Αυτό δεν είναι, επιχείρηση, δεν είναι πρόβλημα της επιχείρησης. Η επιχείρηση ακολουθεί τη φυσική λογική για την οποία έγινε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσει η πολιτική. Την ε, εδαφική διαφορά την κάνει ή με νέο PSU, νέους φόρους δηλαδή, ή με την επιδότηση των υπηρεσιών. Δεύτερο θέμα. Τι πρέπει να υπάρχει κατά βάση. Το πρώτο θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις δραστηριότητες που δίνουν κέρδη και τις δραστηριότητες που έχουν ζημίες. Τώρα, για το αν έχουμε τέντερ ή ανάθεση, δεν σας το, δεν σας το αποφασίσω εγώ. Εμείς σε κάποιες περιπτώσεις διαγωνισμού στην Ιταλία δεν θα μετάσχουμε ή δεν δεχθούμε PSO που ετοιμάζουν ορισμένες ε, περιφέρειες. Γιατί δεν υπάρχει βεβαιότητα πληρωμής και βεβαιότητα κάλυψης του κόστου γιατί να πάμε εμείς ως επιχείρηση πρέπει να σεβαστούμε τους λογαριασμούς επιχείρησης, τα στοιχεία της επιχείρησης. Γιατί να κάνουμε ε, να, να πηγαίνουμε με ζημίες. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών, όχι δικό μας. Το θέμα που έθεσε ο κ. Κανσιάν και άλλοι. Καταρχά, για να επανέλθω και σε, για να, να κτίσουμε αυτό που είπα για, τα εμπο, το, τις εμπορευματικές και τις διεθνείς μεταφορές. Και ισχυρός εθνικός ε, ρυθμιστής και Ευρωπαίος ρυθμιστή Και τι πρέπει να κάνουν. Να θέσουν όλο το πλαίσιο για μια ελεύθερη εγγυημένη πρόσβαση με σαφείς κανόνες, σαφή χρονοδιάγραμμα, σαφές χρονοδιάγραμμα και ισότιμη πρόσβαση όλων. Και εγώ είμαι πεπισμένος ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε στη λογική των εθνικών αγορών. Μία ευρωπαϊκή αγορά θα υπάρχει, όπου επιλέγονται δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Η παλιή συνδεδομική, δηλαδή τρένα, ή η κατασκευαστική βιομηχανία. Και σε μεγάλες επιχειρήσεις θα μείνουν παντού σε αυτές τις αγορές τρεις-τέσσερις επιχειρήσεις. Στον ε, τομέα των, των, των κατασκευαστικών δύο. Οι competitors, οι ανταγωνιστές που έρχονται από την Ιαπωνία και είναι ήδη εδώ, και είναι στην αγορά, είναι το τωρινό πρόβλημα. Κύριε Μωρέτη, τελειώνετε. Τελειώνω. Ισχυρός ρυθμιστής, άνοιγμα της αγοράς γιατί είναι στο διεθνή τομέα, γιατί είναι το 80%. Νέοι κανόνες διατροπικότητας των εμπορευμάτων, γιατί εγώ αν είχα ξεκινήσει στην Ιταλία από τις αγγλικές συνθήκες όπου δεν υπάρχει βασικά ε, εμπορευματικές μεταφορές θα είχα τελείως διαφορετική στάση. Τελειώνω, τελείωσα. Μιλάνο, Βενέτσια. No. Μόναχο, Βενετία. Υπάρχουν έξι στάσεις. Κόβεται ο... Try and keep control of this committee. You... Μα πώς θα ελέγξω λοιπόν. Ξέρω αν ξεπερνάτε όλοι το χρόνο σας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, ίσως. Όλοι ε, εκφράζετε επαρκώς το μήνυμά σας, αλλά πρέπει να απαντάτε κιόλας. Ο κύριος Μπάρκλη. Ευχαριστώ πρώτα. Για το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα έγγραφο που θα το στείλω ηλεκτρονικά σε όλους που θα απαντήσει σε πολλές από τις απορίες σας. Ναι, στην αρχή πήγαν άσχημα τα πράγματα, αλλά ήμασταν και οι πρώτοι που απελευθερώσαμε. Τώρα πήραμε τα μαθήματα. Τώρα αυξήθηκε η κυκλοφορία εμπορευμάτων και επιβατών κατά 60% και μειώθηκε το κόστος κατά 50%. Καλά είναι. Πώς έγινε αυτό για τα εμπορεύματα, ο ανταγωνισμός. 7 εταιρείες Και νομίζω ότι αν θέλετε λοιπόν τα στοιχεία από ανεξάρτητη μελέτη υπάρχει ένα έγγραφο της Κομισιόν που το έχω στο φάκελό μου. Ο αριθμός θέσεων εργασίας στους ιδεοδρόμους ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μειώθηκε πολύ από την απελευθέρωση. Μερικές θέσεις μάλιστα αυξήθηκαν οι οδηγοί ας πούμε. Για τον διαχωρισμό θα ήθελα να σας πω ότι έχουν αυξηθεί και τα κέρδη. Το πρόβλημα του διαχωρισμού και της έγκρισης που πρέπει να χορηγείται είναι μεγάλος φραγμός για ολόκληρη την Ευρώπη. Ρωτήσατε αν υποστηρίζουμε μία διευρωπαϊκή διενοσιακή εποπτεία. Αυτό είναι θέμα χρηματοδότησης. Γιατί όχι όμως. Φυσικά πρέπει να υπάρχει και τοπικός έλεγχος των υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Αλλά όσο πιο ενιαίο γίνεται το σύστημα τόσο το καλύτερο. Η σύγκριση με τη Γαλλία είναι κάτι που είναι δύσκολο γιατί στη Γαλλία υπάρχουν πολλοί φραγμοί και γι' αυτό ο όγκος των εμπορευμάτων στη Γαλλία που κυκλοφορούν με τα τρένα μειώθηκε κατά 50% ενώ όπως σας είπα σε εμάς αυξήθηκε 60%. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερες μελέτες ή όχι. Είναι τόσο λίγοι οι ανεξάρτητες εταιρείες που είναι δύσκολο να έχουμε αντικειμενική άποψη. Αλλά αν θέλουμε να υπάρχει ενιαίο σιδηροδρομικό σύστημα, ας είναι όσο το δυνατόν πιο ενοποιημένο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν διαφορές, είναι μικρότερα τα τρένα και το εύρος των γραμμών. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. αυτό είναι τεχνικό θέμα και τεχνολογικό. Αν όμως υπάρχει ενιαίο σύστημα σηματοδότησης ας πούμε είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί έτσι θα εξοικονομηθούν χρήματα και θα έχουμε την ευκαιρία να αυξήσουμε τον όγκο των κυκλοφορούν των εμπορευμάτων. Κυρία Χέμιν, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Τώρα, γιατί κάνουμε αυτό το πακέτο, γιατί συμμετέχουμε. Μιλήσαμε για την ενιαία ε, εσωτερική αγορά. Θέλουμε ενιαίο διαχειριστή υποδομών. Να έχουμε εναρμονισμένη ε, διαχείριση υποδομών. Τώρα, θα υπάρχουν ε, σε τεχνικό επίπεδο διαφορές ε, ή όχι, ε, θα το δούμε. Αλλά τον αν ενιαίος θα πρέπει να κρυθεί με βάση την επιτυχία που θα έχει και η τέταρτη δέσμη. Πρέπει, μπορεί να, μπορεί να χρειαστεί να πάμε πιο μακριά στο μέλλον με αυτό το όραμα. να περάσει από το λοιπόν η πρόταση από το Συμβούλιο και μετά επανερχόμεθα για να το συζητήσουμε στις λεπτομέρειες. Η κυρία Τρίερ. Τα συνδικάτα δεν είναι κατά της ενιαίας σιδηροδρομικής ευρωπαϊκής αγοράς. Ο τρόπος μας ε, απασχολεί. Δεν νομίζουμε ότι ο πλήρης διαχωρισμός ε, επιχείρησης και υποδομών είναι σωστός και δεν νομίζουμε ότι η απελευθέρωση των εθνικών σιδηροδρόμων και επιβατικών εθνικών υπηρεσιών είναι σωστός τρόπος. Πιστεύουμε ότι η διαλειτουργικότητα είναι ο σωστός τρόπος και μάλιστα θα ήταν ο σωστός τρόπος πρώτα να δημιουργηθεί αυτή η διαλειτουργικότητα. Ως συνδικάτα συμβάλαμε σε αυτό. Η δική μας οργάνωση διαπραγματεύτηκε το 2003 με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Εργοδοτών δύο συμφωνίες που ήταν η Συμφωνία Διαλειτουργικότητας Προσωπικού, μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις συνθήκες εργασίας ε, των διακινουμένων εργαζομένων διασυνοριακά που κατέληξε σε Ευρωπαϊκή Οδηγία και από το 2008 εφαρμόστηκε και σε εθνικό επίπεδο. Η άλλη ήταν για το, την άδεια των οδηγών των σειρμών. Τώρα αυτό είναι παράρτημα στην οδηγία, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους ε, οδηγούς, οπότε συμβάλαμε στη διαλειτουργικότητα, συμβάλαμε στη διευκόλυνση των ε, ε, διασυνοριακών εργαζομένων. Τώρα, η απελευθέρωση μακροπρόθεσμα μπορεί να βελτίωνε την κατάσταση των εργαζομένων αλλά γενικά αναγνωρίζεται ότι η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά τους εργαζομένους. Και όπως είπα και πιο πριν, η αναδιάρθρωση λαμβάνει χώρα εδώ και 10-15 χρόνια στο σιδηροδρομικό τομέα και επηρέασε πολύ τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλου. Δεν μπορώ να τις αναφέρω όλες τις επιπτώσεις, ένα όμως θα το πω. Του χρόνου είναι ε, το έτος ε, ασφάλειας ε, και υγιεινής στον τόπο εργασίας και το βασικό σημείο για τους σιδηροδρόμους είναι η αναδιάρθρωση και η ψυχοκοινωνική κίνδυνη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία έχει ήδη διακηρύξει στόχους ε, ό,τι αφορά τους επιβάτες και τους εργαζομένους, η ερώτηση του κυρίου Γκρός είναι αυτή. Νομίζω ότι οι επιβάτες και οι, ε, ε, επιβάτες και εργαζόμενοι έχουν πολλά κοινά να είναι ασφαλείς οι σιδηρόδρομοι και να είναι ποιοτικέ οι υπηρεσίες. Και στα τρένα και στους σταθμούς ε, κάνουν το πάνι σιδηροδρομική να αποφύγουν τις καθυστερήσεις, αλλά αυτή είναι στην πρώτη γραμμή των παραπώνων. Ε, έχουμε λοιπόν πολλά κοινά συμφέροντα. Συγγνώμη που δεν μπαίνω σε μεγαλύτερο βάθος. Κύριε Κράμερ, νομίζω ότι η ελάχιστη μισθή δεν είναι λύση. Η λύση είναι υποχρεωτικές συμφωνίες ποιότητας που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις σιδηροδρομικές εταιρείες. Στη Γερμανία ετοιμάζονται τώρα και νομίζω ότι η γερμανική μέθοδος για να διασφαλίσουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα είναι η νόμοι για την ε, υποχρεωτική συμμόρφωση στι συλλογικέ συμβάσει. Τώρα στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα που μελετά την κατάσταση αυτή τη στιγμή, είμαστε σε αυτή τη φάση δηλαδή και θα επανέλθουμε με πληροφορίε για την κατάσταση στον τομέα. Συγγνώμη που είμαι τόσο βιαστική, αλλά δεν είχα περισσότερο χρόνο. Ο κύριος Ζακό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη Γαλλία η κατάσταση είναι ότι οι επιβάτες βλέπουν όλο και περισσότερο, όλο και συχνότερα να καταργούνται γραμμές που τις θεωρούμε μη αποδοτικές. Όχι μόνο μικρά δρομολόγια, αλλά και ορισμένα δρομολόγια τρένων υψηλή ταχύτητας που λένε ότι έχουν έλλειμμα. Ενώ ταυτόχρονα η, ο γαλλικός ΟΣΕ λέει ότι έχει κέρδη. Εδώ δεν είναι το κλειδί. Δηλαδή, μήπως για να μην υποστεί τον εσωτερικό ανταγωνισμό υφίσταται περισσότερο τον εξωτερικό ανταγωνισμό από άλλους τρόπους μεταφοράς. Αυτό γίνεται για τα εμπορεύματα τουλάχιστον. Και οι εργαζόμενοι υποφέρουν περισσότερο από την εξωτερικό παρά από τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Συχνά ζητούμε να ξανανοίξουν γραμμές, να ανακαινιστούν οι υποδομές και μας λένε δεν έχουμε λεφτά. Αλήθεια μεν είναι, όλοι αυτό το πρόβλημα είχαν ανέκαθεν, αλλά τώρα το ξέρουμε. Για να έχουμε λοιπόν περισσότερη απόδοση με τα χρήματα που διαθέτουμε, χρειάζεται αναδιοργάνωση εσωτερική. Δεν θα σας πω πώς θα γίνει, αυτό θα το κάνει η SNCF, αλλά θα μπορούσε να επιτευχθεί και με μείωση του προσωπικού μεταξύ άλλων. Αυτό το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Τι να προσθέταμε στην τέταρτη δέσμη. Εδώ είναι θέμα των λεπτομεριών δηλαδή. Να σταματήσουμε να ζητάμε καλύτερο συντονισμό. Ζητάμε μάλλον συνεχώς ε, καλύτερο συντονισμό μεταξύ οργανώσεων επιχειρηματιών και επιβατών. Θέλουμε να μας ακούσουν για την ποιότητα των υπηρεσιών και της πληροφόρησης. Σας το είπα και πριν. Για την ποιότητα για τη χορήγηση των εισιτηρίων, την έκδοση των εισιτηρίων που γίνεται όλο και περισσότερο από μηχανές και ίντερνετ ενώ δεν μπορούν πολλοί να χρησιμοποιήσουν τους τρόπους αυτούς. Να, ορισμένες ιδέες για καλύτερη συντονισμό και συνεργασία. Έγινε πολλής λόγος για το διαχωρισμό των διαφόρων οργανισμών που θα διαχειρίζονται τις υποδομές κτλ. Μετα, μάλλον διαχωρισμό μεταξύ διαχείρισης των υποδομών και επιχείρησης των σιδηροδρόμων. Αλλά χρειάζεται συνεργασία, όχι μόνο διαχωρισμός, γιατί να μην υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ οργανισμών που νομικά θα είναι χωριστή. Στη Δανία έχω δει να συνυπάρχουν στην ίδια αίθουσα οι διαχειριστές των υποδομών με τους διαχειριστές των τρένων. Είναι δυνατή η συνεργασία και έτσι λύνονται αυτόματα τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση του κυρίου Γκρός, αν μπορούμε να ελέγχουμε τις οικονομικές, τις χρηματικές ροές, όχι, όχι όπως το εννοείται. Μπορούμε να ελέγξουμε τις ε, ροές αυτές ε, όταν οδηγούν σε διακρίσεις ε, σε κάποιες περιφέρειες όπου οι τιμές ήταν ψηλέ λόγω ανταγωνισμού. Αν... Εμείς είμαστε κατά των διεπιδοτήσεων ε, που στηρίζονται σε τέτοια συστήματα εταιριών συμμετοχών. Κύριε Καρδούη, καταλαβαίνετε ότι δεν υπερασπίζουμε το γερμανικό μοντέλο καθ' ολοκληρίαν. Ναι, εγώ θέλω ρεαλιστικά να δούμε τα προβλήματα και αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει θεωρητική για το unbundling και το διαχωρισμό να την αφήσουμε κατά μέρος. Πολλά μπορούμε να βελτιώσουμε στους σιδηροδρόμους. Έχουμε τώρα ένα νόμο που συζητείται στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και θα συμμετέχω την επόμενη Τετάρτη σε μια ακρόαση. Πρόκειται για την περαιτέρω ενίσχυση της ρυθμιστικής αρχής. Πρέπει οι τιμές από, ε, από την αρχή εκ των προτέρων να εγκρίνονται. Επίσης θα ε, υπάρξουν... Ε, και άλλες συζητήσεις ε, για τις διακρίσεις κλπ. Όλα αυτά θα τα ε, ε, τακτοποιήσει ο καινούριο νόμος. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να βελτιωθεί ακόμα το γερμανικό σύστημα και προσθέτω ότι οι διάδρομοι, τρεις περνούν από τη Γερμανία και οι διάδρομοι αυτοί θα είναι μια δοκιμία ας πούμε, θα είναι η Λιδία και θα δούμε εάν και οι τοπικές μεταφορές θα λειτουργούν καλά και αν οι τιμές θα είναι σε σωστό επίπεδο. Ε, δεν νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα ε, αναθέσουμε σε έναν Ευρωπαίο ε, ρυθμιστικό φορέα. Ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση, με την παράδοση που υπάρχει στις ε, υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και αυτό ισχύει για τη Γερμανία. Ε, πολλές φορές ε, όλα αυτά οδηγούν σε βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους επιβάτες. Μιλάμε λοιπόν για εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς. Αν υπάρχουν προβλήματα υπάρχει και η δικαστική προσφυγή. Ε, νομίζω ότι στους, στις τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχει, ούτε στην ενέργεια υπάρχει ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας. Άρα δεν χρειάζεται νομίζω καταρχήν στους σιδηροδρόμους. Ας έχουμε τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς. Εγώ διαπιστώνω ότι ε, οι υπηρεσίες παρέχονται από κατεστημένους φορείς εκμετάλλευσης μόνο ε, θέλετε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός ε, με το σωστό τρόπο εάν το επιχειρήσετε θα συνεργαστούμε και εμείς. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν ζήτησε το λόγο. Έχουμε τρία λεπτά. Κυρία Μπράουτη, άμα θέλετε να μιλήσετε τώρα. Πρέπει να τελειώσουμε στις 12.30. Όλοι μίλησαν για τα δικαιώματα των εργαζομένων, υπάρχουν και τα δικαιώματα των διαρμηνέων Και το ωράριό του προβλέπεται να διακοπεί στι 12.30 Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και μα δίνετε, που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Θα είμαι πολύ σύντομη. Πρώτον, για τον, ε, την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή. Το κείμενο της αναδιατύπωσης έχει σαφή ρήτρα να υποβάλει έκθεση η Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή, θα το κάνουμε. Έγιναν σχόλια για το κατά πόσον είναι ή όχι αναγκαίο το πακέτο. Όπως ξέρετε, και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις και όπως είπε η κυρία Χάιμινγκ, καλύπτει ένα σαφές κενό που απαιτεί νομοθετική κάλυψη. Μετά έγιναν σχόλια για την, τον, τη μελέτη αντικτύπου και αν είναι παρκώς παρασκευασμένο το κείμενο. Σας διαβεβαιώ πως ναι. Η Επιτροπή έχει ετοιμάσει τρεις μελέτες αντικτύπου με πολύ ε, ε, ξεκάθαρο και ε, αυστηρό τρόπο έχοντας διαβουλευθεί τους, ε, όλους τους φορείς, κάτι που δεν, είναι ακρίβη, που δεν συμβαίνει στις μελέτες που ετοίμασε η CER και άλλοι Πιστεύουμε ότι η μελέτη αντικτύπου είναι απόλυτα διαφανής και ως προς τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσει, και αν θέλετε να ενημερώσουμε τους ε, ε, βουλευτές για, τον αντικ... για, τη μελέτη για τις μελέτες αυτές όποτε θέλετε. Για την ανάγκη ισχυρού ρυθμιστή, ρυθμιστική ρυθμιστικής αρχής. Ναι, η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι αρκετή. Υπάρχουν, ξεκίνησαν, ξεκινούν Οχτώ νέε διαδικασίε ε, από τι υφιστάμενε αρχέ για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση, η ισότιμη πρόσβαση. Όπως αναφέρεται αυτό απαιτεί τεράστιο κόστο ε, και, σε, οικονομικό και σε χρόνο. Πώς οι νέοι εισερχόμενοι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή για να μπουν στην αγορά. Ευχαριστώ. Στο, στις 12.30 just σταματάμε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, τους βουλευτές επίσης. Ζητώ συγγνώμη που ήμουν ομός απέναντι, βάναυσος απέναντί σας. Ξέρω ότι έχω τη φήμη του βάναυσου, όντως έτσι είναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι τελειώσαμε έγκαιρα και ως υπεύθυνοι των σιδεδόμων ξέρετε ότι όταν κανείς φτάνει στην ώρα του είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα τρένα. Θα τα πούμε το απόγευμα στις 3 για το δεύτερο τμήμα συζητήσεων. Ευχαριστούμε. Καλή σας όρεξη.